Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε, ούτως ώστε χωρίς να καθυστερήσουμε πολύ περισσότερο, να μπορέσουμε να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Σημείο 1 ε, για την έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης ε, θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουμε αλλάξει τη σειρά στο, στα σημεία που θα εξετάσουμε, τα σημεία 7 και 14, ε, τροπολογίες και εξέταση σχεδίου έκθεσης της κυρίας Μάκιντάιρ αναβάλλονται για την συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στις 23 και 24 Ιανουαρίου. Το σημείο 25, εξέταση τροπολογιών της έκθεσης του κυρίου Γκοτιέρο, αναβάλλονται για την έκτατη συνεδρίαση της Επιτροπής μας σε 9 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια μετά το σημείο 27 προστίθεται και άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη 27 Α για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ως προς την ε, διεξαγωγή έρευνας για την αγορά σε ε, έκθεση Αντοκά. Και τελευταίο σημείο, πρόοδος για τις διαπραγματεύσεις για την οδηγία σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Πρόκειται ε, για την Ταλότα ζοβιέσκα επίσης. Ε, αν δεν έχετε ενστάσεις, θεωρώ ότι εγκρίνονται αυτά τα σημεία. Έχω και τέσσερις ανακοινώσεις να σας κάνω. Πρώτον, θέλω να σας θυμίσω ότι μετά τις εργασίες μας σήμερα το απόγευμα θα κάνουμε ένα κοκτέιλ για το τέλος του έτους για το καλό. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ, είστε όλοι ευπρόσδεκτοι σε κάθε περίπτωση. Ε, για να ευχηθούμε όλοι σε όλους ε, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Ε, ως προς την επόμενη συνεδρίαση, 23 και 24 Ιανουαρίου, θα ήθελα να σας πω ότι το απόγευμα της 23ης ακυρώνεται η συνεδρίαση. Στις 12.30 θα ε, είστε ελεύθεροι λοιπόν, εκτός ε, βεβαίως ε, από όσους μετέχουν στον τριμερή διάλογο για την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Euh, ε, ένα σημείο που επανέρχεται διαρκώς, το θέμα δηλαδή της διερμηνίας όταν δεν γίνεται χρήση των υπηρεσιών διερμηνίας, λυπάμαι ε, που θα σας πω πως πρέπει να ε, πραγματευτούμε σοβαρά αυτό το σημείο, διότι η ισπανική ε, διερμηνία δεν χρησιμοποιήθηκε στην ε, πλειονότητα των συσκέψεων των σκιωδών για την έκθεση Μάκιντερ, διότι ο σκιώδης από σοσιαλιστές, ο κύριος Σέζιο Γκουτιέρες, παρευρέθη σε πολύ μικρό μέρος της συνεδρίασης των σκιωδών. Τέλος, για ε, το προγραμματισμό των εργασιών μας ε, μπορείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις στο ίντρανε, το εσωτερικό ε, δίκτυο. τι άλλο, να σας πω ότι έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, ενστάσεις, οτιδήποτε, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα με το πέρας της συνεδρίασης. Σημείο ο κύριος Κάσλερ δεν είναι εδώ. Τι θα κάνουμε τώρα. Ο κύριος Ντεμπάκερ επίσης απουσιάζει. Ούτε ο κύριος Κάζα είναι εδώ. Η ε, υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για αυτούς τους βουλευτές να κάνουν τα απαραίτητα ε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε νωρίτερα τις ψηφοφορίες. On me dit que le, le groupe Μου λένε ότι το ΕΛΚ έχει καταφέρει να επαναφέρει τα πράγματα σε τάξη. Από πλευράς των φιλελευθέρων υπάρχουν νέα. Ο κύριος ε, Ντεμπάκερ ε, θα έρθει το ταχύτερο δυνατόν as soon as possible, όπως λένε και οι Γάλλοι όταν μιλάνε αγγλικά. Bien, dans la course, c'est les libéraux qui l'ont emporté. Ε, κέρδισαν στον αγώνα δρόμο, οι φιλελεύθεροι. Νίκησαν και το ΕΛΚ. Ε, τους πρόλαβαν και θα αρχίσουμε με το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Ε, τι να πω τώρα για τα μέλη του ΕΛΚ που είναι εδώ πέρα. Ε, προς, προς σημείο 5 λοιπόν. Εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών για την έκθεση Ντεμπάκερ. Πρόκειται για την έκθεση Επιτροπή Μεταφορών για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. Εκδίδουμε χνομοδότηση με αποδέκτη την Επιτροπή Μεταφορών και ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Φιλίπ Ντεμπάκερ. Οκτώ συμβαστικές ε, τροπολογίες έχουν συνταχθεί. Δίνω το λόγο στον εισαγητή. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που άργησα. Ναι, πρέπει να συζητήσουμε τι συμβαστικέ τροπολογίε τη γνωμοδότηση αυτή για τον κανονισμό όσον αφορά την ε, ε, πολιτική μα για λιμένες και λιμενικές υπηρεσίε. Έγινε πολύ επικοδομητική η συνεργασία μα όσον αφορά εμένα και μεταξύ μου τόσο πάνω και των σχεδόν συζητών των πολιτικών ομάδων και προσπαθήσαμε, όπως προσπάθησε δύο φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περάσει την πρότασή της, είναι η τρίτη. Και, όπως λέμε, τρίτη και φαρμακερή. Ας ελπίσουμε ομένως ότι αυτή τη φορά όντως θα το πετύχουμε. Επομένως, ε, καταλήξαμε σε αυτούς τους οκτώ, οκτώ συμβαστικές τροπολογίες, όπως προείπα, και να σας πω τα πρώτα πρώτα το ιστορικό πλαίσιο όσον αφορά τους συμβασμούς για τα σχετικά άρθρα. Άρθρο 10, παράγραφος 2. Εδώ ε, τα κράτη-μέλη ε, υποχρεούνται να εφαρμόσουν ε, τις λιμενικές αρχές να σεβαστούν την οδηγία 2023. Το ε είναι μια μικρή αλλαγή σε σχέση με το άρθρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μετά έχουμε το D ε, και λέμε εδώ πέρα ότι θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση των λιμενικών αρχών προς την νομοθεσία για τα κοινωνικά μέτρα και είπαμε ότι θα πρέπει να διαβουλεύονται με τους εργαζομένους οι λιμενικές αρχές και είπαμε ότι και αυτό είναι βελτίωση τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα για τι παραγράφου και εδώ έχουμε κάποιε τέτοιε ε, σωστικέ τροπολογίε και επιφέρουμε και τι Έχουμε όμω δύο προφορικέ τροπολογίε από τον κύριο Χάουι Κατά τη γνώμη μου, ε, δεν ταιριάζουν για το έγραφο 8 πράγμα 6 εδώ θα προτιμούσα αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορώ να συμφωνήσω με την πρόταση όμως του κυρίου Μπαχ διότι θεωρώ ότι εδώ ε, υπάρχει παραπομπή στο άρθρο 28 της συνδίκης και η προφορική τροπολογία όπως έχει σήμερα ε, δεν με βρίσκει σύμφωνα ούτε εμένα, ούτε την πολιτική ομάδα, αλλά ούτε και άλλε πολιτικέ ομάδε. Θεωρούμε ότι πάει πολύ, είναι υπερβολική τέλο πάντων. Ε, άρθρα 17 και 18 και εδώ έχουν συμφασικέ τροπολογίε. είπαμε όμως ότι είναι απαράδεκτε γιατί αφορούν ε, δεν αφορούν τους πάντων και είπαμε ε, να διαγραφούν το είπε ο και γι' αυτό έχουμε την προφορική τροπολογία είναι μια μικρή μεταβολή τώρα όμω, επειδή κηρύχθηκαν απαράδεκτε, μπορούμε να δούμε τι θα πει η Επιτροπή Μεταφορών γιατί και εκεί συζητείται το θέμα Οπότε να δούμε τελικά αυτή η δεσμή μέτρων που θα καταλήξει και τι θα γίνει με τι εποπτικέ αρχέ των κρατών μελών. Και έτσι να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων. Ελπίζω και ο κύριο Χάβιτ να συμφωνήσει. Uh, direct. Κάτι άλλο επίσης όσον αφορά την οδηγία για τις εκχωρήσεις, αδειοδοτήσεις. Ε, έχουμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο επιδέχεται βελτιώσεις. Αλλά ούτε αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας ως Επιτροπή Απασχόλησης. Έχει να κάνει με τις μεταφορές και υπάρχει άλλη οδηγία, πιο ειδική. Και πήγα και γύρω στην Ευρώπη σε έξι λιμένες. Η κάθε λιμενική αρχή έχει άλλη ερμηνεία για αυτή την ε, οδηγία. Και γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να ζητηθεί αυτό το θέμα όχι μόνο σε σχέση με την απασχόληση, αλλά ευρύτερα, γενικότερα. Επομένως, αυτά για όλα αυτά τα δύσκολα ζητήματα. Πολλοί φοβόντουσαν ότι δεν θα καταλήξει καλά αυτή η ιστορία. Όμως, ήταν θετική συνεργασία με όλους τους σκιώδεις ηγητές. Γι' αυτό και καταλήψαμε σε αυτούς τους πετυχημένους συμβιβασμούς. Τώρα νομίζω ότι αυτή η γνωμοδότηση μπορεί να είναι μια σωστή αφετηρία για τη δουλειά μας και για τη δουλειά της Επιτροπής των Μεταφορών και θα δούμε και θα αποδειχθεί όταν γίνει ψηφορία σήμερα ότι καλύπτουμε αυτά τα οποία θέλαμε και λοιπόν θα δοθεί και αίσια συνέχεια και στην Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε και τώρα Στην του Μπαχ η κυρία Σαγιάκη. Αγαπητοί συνάδελφοι, Δυστυχώ, ο κύριος Μπακ ε, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα γιατί ε, είναι στην Επιτροπή Μεταφορών όπου είναι απαραίτητος για την ε, υπερψήφιση της έκθεσής του. Μου ζήτησε λοιπόν να διαβάσω εκ μέρους του ονόματός του τη δήλωσή του. Ευχαριστεί τον εισηγητή και τους εισηγητές για την πολύ καλή συνεργασία και για τις συζητήσεις που έγιναν ανάμεσά τους. Ε, λόγω της μεγάλης ιστορίας και της ευαισθησίας αυτού του φακέλου της υπόθεσης αυτής. Δεν ήταν εύκολο να υπάρξει συμφωνία, αλλά ελπίζει να υπάρξει καλό σημασμό στα περισσότερα θέματα. Επιθυμεί να εκφράσει την υποστήριξή του για όλες τις συμβαστικές τροπολογίες, να και στηρίζει την πλειοψηφία των τροπολογιών. Επίσης χαίρεται που καταλήγουμε σε συμφωνία όσον αφορά το EA. Οι σοσιαλιστές συμφωνούν, μισό λεπτό, συμφωνούν με το A και DA με αυτές τις τροπολογίες. Επιπρόσθετα στηρίζει την προφορική τροπολογία του κυρίου Χάουιτ για τη δική του την τροπολογία 56 που αφορά ε, στο άρθρο 8 παράγραφος 6. Ε, το θέμα αυτό είναι λιγάκι επίμαχο και με βάση αυτά που είπε ο εισηγητής, αλλά θα γνωρίζετε ήδη ότι υποστηρίζει αυτή την προφορική τροπολογία. Αυτά λοιπόν είναι τα σχόλια του κυρίου Μπάκα, το τι επιθυμεί και του κυρίου Μπάκα ευχαριστεί για τη συνεργασία. Richard Uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καταρχήν ε, θέλω να πω ότι ευχαριστώ τον κύριο Μπάκα ε, γιατί έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Νομίζω η δυσκολία που υπάρχει είναι ότι υπάρχει διάσταση απόψεων και νομίζω ότι έκανε ό,τι μπορούσε έχοντας κατά νου αυτή τη διάσταση των απόψεων. Έχουμε σημειώσει αρκετή πρόοδο και θέλω να τον ευχαριστήσω και να τον συγχαρώ. Όσον αφορά λοιπόν ε, διότι έχει ε, αποκαλέσει, έχει μιλήσει και για κόκκινες γραμμές. Εμένα δεν μου αρέσει να κάνουμε ε, χρήση τέτοιου είδους ε, διατυπώσεων, προτιμώ να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Όσον αφορά την πρόταση απόρριψης, εμείς θα υπερψηφίσουμε και αυτό θα το κάνουμε γιατί ε, υπάρχουν πολλοί που εκπροσωπούν τον κλάδο και τους λιμένες και θέλω να επαναλάβω αυτό που έχω ξαναπεί και στις διαπραγματεύσεις, ότι εμείς εμείς ε, διαπραγματευτήκαμε χωρίς ε, προκαταλήξεις για να καταλήξουμε στη βέλτιστη δυνατή λύση και παραμένουμε στις συμφωνίες μας. Πάντως, ε, όπως σας είπα, εμείς θα υπερψηφίσουμε και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ανάλογα θα συμπεριφερθεί και η Επιτροπή. Και κάτι άλλο να πω. Είμαι αρκετά ευτυχής που μπορώ να επιβεβαιώσω ότι στηρίζουμε τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Όσον αφορά κυρίως το 16, ε, θέλω να σας πω ότι ήμασταν σε θέση να καταλήξουμε σε συμφωνία σε αυτό το τόσο δύσκολο θέμα ε, του τι θα προέκυπτε εάν υπήρχαν συλλογικές διαμαρτυρίες να σας πω ότι πραγματικά είναι απογοητευτικό το ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε επί του άρθρου. Και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ΕΛΚ έχει αφήσει ανοηθεί ότι είναι πρόθυμοι να δεχτούν την προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών για το άρθρο A. Ε, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ντεμπάκερ κατά πόσον και εκείνο ε, ε, θα μπορούσε να συμφωνήσει έτσι ώστε να περάσει αυτή η τροπολογία γιατί θα μπορούσε κανείς ε, να στηρίξει αυτή την τροπολογία και αργότερα. Ε, σας είπα, οι κόκκινες γραμμές δεν μου αρέσουν αυτές οι διατυπώσεις. Ε, αναφέρομαι στην ε, παράγραφο 28 για τις υπεργολαβίες. Είχαμε εδώ μια μακρά συζήτηση και πραγματικά υπάρχει ουσιαστική διάσταση απόψεων. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εάν λοιπόν η δική μας η τροπολογία δεν περάσει, τότε αυτό σίγουρα θα πειράσει το τελικό κείμενο. Εάν λοιπόν θέλει να συζητήσουμε γι' αυτό, τότε οπωσδήποτε θα αλλάξει η θέση των σοσιαλιστών και των δημοκρατικών, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά σε αυτή την Επιτροπή που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της υπεργολαβίας. Αυτός είναι ένας τρόπος για να αποφύγει κανείς την κοινωνική προστασία και κατά την άποψή μου ισχύει στην περίπτωσή μας αυτό. Εάν λοιπόν ε, δεν ε, στηριχθεί η απόρριψη. Εμείς θέλουμε να περάσουν αυτές οι τροπολογίες. Χαίρομαι πάρα πολύ, εν που υπήρξαν όλοι αυτοί οι συμβασμοί και εμείς ε, τηρούμε τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί. Η κυρία Σουρούντερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια, εδώ πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, γιατί εδώ δεν πρόκειται μόνο για λιμενικές υπηρεσίες, πρόκειται κυρίως ε, και για το πώς θα ρυθμίζονται αυτές, με πιο εργατικό δίκαιο και κατά πόσον ε, θα υπάρχει πίεση ε, σε σχέση με το ισχύον δίκαιο στα λιμάνια. Θυμόμαστε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι υπήρξαν μεγάλες διαδηλώσεις, εδώ μάλιστα στο Κοινοβούλιο, όπου ελέγχθη ότι αν τελικά δεν βρείτε μία δίκαιη λύση, τότε ασκήθηκε μάλιστα κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ε, είναι σε μία φάση που ε, αποδυναμώνει τις ε, προδιαγραφές ασφαλείας. Σήμερα λοιπόν φέρουμε τεράστια ευθύνη. Πράγματι έχει δίκιο ο εισηγητής ότι είχαμε καλές διαπραγματεύσεις, επιτύχαμε αρκετά και μάλιστα συνεχίζουμε σε κάποιο βαθμό αυτά τα οποία προσπάθησαν να ε, συνεχίσουν οι κοινωνικοί εταίροι, να βρούμε δηλαδή μια εξισορροπημένη στάση. Επίσης ε, υποστηρίζουμε ε, τους κεντρικούς συμβιβασμού, διότι ο εισηγητής ήρθε και αυτός προς εμάς. Στηρίζουμε λοιπόν τους περισσότερους συμβιβασμού, αλλά θεωρώ ότι είναι προβληματικό και το λέω αυτό με απόλυτη σαφήνεια όταν μία παράγραφος έρχεται μετά από ένα συμβασμό στο αμέσως επόμενο άρθρο όπου με αυτή την προστίκη εξαφανίζεται ο συμβασμός. Αναφέρομαι στον συμβιβασμό DA για το 4 παράγραφος 2 σημείο DA. Και αμέσως μετά στο 4-3... λέμε ακριβώς το αντίθετο αυτού που έχει επιτευχθεί στο συμβιβασμό. Δηλαδή λέμε ότι υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές και μετά όμως αναφέρεται ότι είναι περιορισμένες αυτές οι προδιαγραφές. Άρα δηλαδή όλα αυτά που έχουμε πετύχει διαλύονται. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε κατά πόσον ένα τέτοιο άρθρο καταπίπτει όταν λέει ακριβώς το αντίθετο. Για μας λοιπόν τους πράσινους αυτό είναι καθοριστική σημασία. Γιατί αν με τον τρόπο αυτό έρεται η συμβαστική πρόταση, εμείς δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε. Για μας λοιπόν τίθεται το ερώτημα κατά πόσον η τροπολογία 44 δεν καταπίπτει εφόσον υπάρχει η συμβαστική πρόταση. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί. Και στην περίπτωση που το άρθρο 44 περάσει, γιατί ο εισηγητής έχει δώσει θετικό πρόσημο, τότε ε, να υπερψηφίσουμε γιατί ε, δεν θέλουμε να καταστραφεί αυτό ε, για το, το οποίο επιτύχαμε μέσα από εργόντις προσπάθειες. Φαντάζομαι ότι δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Θα ακούσουμε τον εισηγητή για να μας απαντήσει μεταξύ άλλων σε αυτήν την τελευταία παρέμβαση, γιατί από ό,τι κατάλαβα του ευθύνατε μια ερώτηση για την, τον κατάλογο ψηφοφορίας. Ε, πρόεδρε, εξαπνιάζομαι και είμαι και λίγο απογοητευμένος, ομολογώ. Ε, πολλές ε, ώρες ε, εργαστήκαμε μαζί μέσα σε ένα πολύ επικοδομητικό πνεύμα και καταφέραμε να καταλήξουμε σε αρκετά καλές συμβαστικές λύσεις. Πολλές πολιτικές ομάδες είπαν ότι δεν θέλουν να διαπραγματεύονται με κόκκινες γραμμές, με απριόρι και προβλήματα και προκαταλήψεις κτλ. Ε, τώρα μισή ώρα, μία ώρα, δύο ώρες πριν από την ψηφοφορία, ε, τι, αντιφάσκουν ε, οι συνάδελφοι. Γι' αυτό και εγώ απογοητεύτηκα. Προσπαθήσαμε να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή και έγιναν ιδεολογικού χαρακτήρα συζητήσεις μεταξύ άλλων. Όμως πιστεύω ότι με τη διατύπωση στην οποία καταλήξαμε και βελτιώσαμε την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρήκαμε μια εξισορροπημένη λύση που θα διαβάσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών καθώς και μια καλή βάση για τις μελλοντικέ μας συζητήσεις. Ε, στην πρώτη παρέμβαση σας είπα ότι όταν συναντιόμασταν με τους σκιώδες συνειδητοποιήσαμε ότι ε, οι περισσότερες αρμοδιότητες Επιτροπής Μεταφορών ε, ε, παρεκτράπησαν προς τον κοινωνικό διάλογο ηθελημένα κατόπιν αιτήματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγώ στην ανακτήρια παρέμβασή μου είπαμε ας του δώσουμε μια ευκαιρία, ας διαπραγματευτούμε ανοιχτά και ας δώσουμε μια ευκαιρία στον κοινωνικό διάλογο και ρητά το αναφέρουμε. Λέμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε να ε, επιτρέψουμε στον κοινωνικό διάλογο να δώσουμε μια ευκαιρία ούτω ώστε να λύσουμε τα προβλήματα που είχαμε στα δύο πρώτα πακέτα για τους λιμένες. Δεν θέλουμε να παραφορτώσουμε αυτήν την ε, γνωμοδότηση ε, και κατά τη γνώμη μου υπάρχουν παράλογες κόκκινες γραμμές. Είναι σημαντική η πρόοδος που έχουμε κάνει και μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τις συζητήσεις μας με την Επιτροπή Μεταφορών. Για μένα Ξέρω, ο κύριος Χάουιτ και πάντοτε το έλεγε και στην πράξη κάναμε μια πραγματικά ανοιχτή συζήτηση για όλες τις συμβαστικές και μας λέει ότι τι θα αρχίσουμε με ε, αρνητική ψηφοφορία ή θετική ψηφοφορία για την τροπολογία που απορρίπτει όλες τις υπόλοιπες. Δεν καταλαβαίνω, τόσες ώρες δουλεύαμε με τους συναδέλφους και τώρα θα, ε, θα ε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Επιλογή σας είναι, κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά πάντως έχουμε ε, κάνει πολλές υποχωρήσεις για να ε, σας ικανοποιήσουμε. Όλοι δώσαν, υποχώρησαν, είναι εξισορροπημένη η λύση. Τώρα τι, ε, ε, νομίζω ότι είναι παράλογο να απορρίψουμε την γνωμοδότηση εξ ολοκλήρου και άρα και την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 8-6. Αρχικά ε, ασχολιόμασταν σχεδόν αποκλειστικά με την τροπολογία ε, και εγώ δέχτηκα να απομακρυνθούμε από τη θέση τη δική μου και της ομάδας. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο ιδεολογικό χάσμα. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό και πρέπει να το σεβαστούμε ε, και είναι και μόνο η λογική προσέγγιση που μπορούσαμε να υιοθετήσουμε. Αυτά ε, είναι τα σχόλια που μπορώ να κάνω. Ελπίζω να το σκεφτείτε σοβαρά διότι ακολουθούμε ε, τη σωστή κατεύθυνση και στις ομάδες σας μπορείτε να το αιτιολογήσετε και να πείτε ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση και έτσι μπορούμε να διασκεδάσουμε τους φόβους ε, που υπάρχουν σε σχέση με την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθήσαμε ε, μέσα σε ανοιχτό πνεύμα να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι το ξέρετε και νομίζω ότι αν ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή στην ψηφοφορία ε, θα μπορέσουμε στις μελλοντικέ συζητήσει με την Επιτροπή Μεταφορών να σημειώσουμε ε, περαιτέρω πρόοδο και να έχουμε καλή έκβαση στην ψηφοφορία. Πρόεδρος, ε, ευχαριστούμε κύριε Σιγητά και παρά την απογοήτευσή σας θα δούμε τη μελγενέστε στην ψηφοφορία, δεν θα αργήσει. Στο μεταξύ μπόρεσε να έρθει ο κύριο Κάσλερ ή εξαφανίστηκε και πάλι. σας προτείνω να πάμε στο σημείο 4 για να εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες ε, για τη γνωμοδότηση που έχει συντάξει ε, με αποδέκτη την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για το πρόγραμμα Solvit. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κέσλερ για να μας ε, παρουσιάσει τις συμβαστικές τροπολογίες. Κύριε Σιγητά. Σας Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που καθυστέρησα. Ήμουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντο. Ε, δεν είχα δει στη μέση διάταξη ότι είμαι πρώτο. Σα ευχαριστώ πολύ που δείχνετε κατανόηση στις συμβαστικές προτάσεις που στηρίζονται από πέντε πολιτικές ομάδες κατ' ουσίαν ε, καλύπτουμε όλες τις επιθυμίες επειδή είναι λίγο πριν από τα Χριστούγεννα γι' αυτό και στο προβληματικό αυτό θέμα του Solvit κατορθώσαμε να ικανοποιήσουμε σχεδόν όλους γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναντέλφους των σοσιαλιστών, των πρασίνων ε, των φιλελευθέρων ε, των συντηρητικών μεταρρυθμιστών το έγγραφο οποίο καταλήγουμε είναι πάρα πολύ καλό. Στην πρώτη ε, συμβαστική πρόταση θέλω να σας ε, επισημαίνουμε πώς μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά το Solvit ε, σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Εδώ έχουμε βελτιώσει κατά τη μία πρόταση που δεν υπήρχε στο προηγούμενο σχέδιο. Στο τέλος, ε, κάτι που θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα είναι μία ε, τροπολογία, ε, τρίτη τροπολογία και εκεί αναφέρουμε και πάλι το ρόλο των εθνικών θεσμών. Θα πρέπει να υπάρχει μια κεντρική έδρα για το Solvit, κεντρική διαχείριση του θέματος και πρέπει να μεριμνήσουμε οι υπηρεσίες Solvit να μπορούν να βοηθήσουν και σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή να βρίσκονται και στην πρωτεύουσα μιας χώρας, αλλά και σε μικρότερες περιφέρειες. Τέλος, Αν δει κανεί τον κατάλογο ψηφοφορία, σχεδόν σε όλα τα σημεία υπάρχει θετικό πρόσημο. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μακρηγορήσουμε. Ε, θα πρέπει να ψηφίσουμε ταχύτατα ε, και ελπίζω να μεριμνήσουμε το Solvit να είναι πιο ορατό, ε, οι άνθρωποι πόσων έχουν προβλήματα ε, με την ομοθεσία της Ευρώπης να μπορούν να στραφούν σε αυτό. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που στηρίζετε κι εσείς αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Θα ήθελαν κάποιοι συνάδελφοι το λόγο, παρακαλώ. Ε, Μπαλτατσίνο. Ε, Ο Ακούσαμε με προσοχή τον εισηγητή και όντως πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Εάν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα στις σχέσεις τους με, τις, ε, με τη διοίκηση, όχι σε μόνο σε επίπεδο ε, κράτους μέλους αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χρειάζεται ένας ε, μηχανισμός για να επιλύονται αυτές οι διαφορές με αποτελεσματικό τρόπο. Χαιρόμαστε λοιπόν που ε, συμμετέχουμε στην εγκαθίδρυση ενός ε, τέτοιου μηχανισμού ε, καταθέντως τροπολογίες. Θέλουμε να ενισχυθεί η λειτουργία αυτού του μηχανισμού Solvit όχι μόνο προβάλλοντας τον περισσότερο δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο. Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Ένα εργαλείο χάρη στο οποίο ε, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λύνουν ε, ταχύτερα τα προβλήματα που έχουν στη σχέση τους με τη διοίκηση. Αυτό το εργαλείο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο και για, τους, ε, για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες, ε, διότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υφίστανται διακριτική μεταχείριση ε, θα χρειαστεί επίσης να προβάλλουμε αυτό το εργαλείο σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Ελπίζουμε λοιπόν να είναι επωφελής αυτή η υπηρεσία για όλους τους πολίτες της Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Ο κύριο Κέσλερ δεν θέλει πάλι το λόγο. Θα ψηφίσουμε λίγο αργότερα. Φτάνουμε εσύ ως το σημείο 6 γνωμοδότηση που εκδίδουμε για τις επιτροπές περιβάλλοντος και βιομηχανίας. Είναι οι δύο συνδεδεμένες επιτροπές για μια γνωμοδότηση ιδίας πρωτοβουλίας με στόχο την, ε, τον ορισμό Ενό πλαισίου για την ενεργειακή πολιτική και την πολιτική για το κλίμα με ορίζοντα το 2030. Η γνωμοδότησή μα ε, συνετάχθη υπό την αιγίδα του κυρίου Κάζα και θα του δώσω το λόγο για να μα παρουσιάσει τι συμβαστικέ τροπολογίε ε, που έχει συντάξει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προσπάθησα στο μέτρο του δυνατού να αποδώσω όσο γίνεται περισσότερο τη σημασία που έχει αυτό το θέμα στην έκθεση και πρόκειται εδώ πέρα για το εργατικό δυναμικό και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται ε, στα θέματα απασχόληση σχέση με την κλιματική αλλαγή. Δεν θα με κατηγορήσω κύριε Πρόεδρε, δεν θα με κατηγορήσω γιατί κατάφερα ε, να καταλήξω σε πέντε συμβατικές τροπολογίες με τους εμπλεκομένους. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό οι δεξιότητες των εργαζομένων εδώ να τονιστούν και αυτό να τονιστεί σε σχέση με τις ανάγκες της ε, βιομηχανίας μας. Ε, εντάξει, φτάσαμε κοντά στις διακοπές, οπότε τελικά πρετάνευσε το μνήμα των Χριστουγέννων και καταφέραμε να κλείσουμε το θέμα. Θα γίνει και ψηφοφορία θα πρέπει τους συναδέλφους όλους, ε, τον Τιβέδη, τον Λάμπερ και όλους, ε, να τους ευχαριστήσω διότι χωρίς τη βοήθειά τους δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποιες σε αυτούς τις διατάξεις. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, Πρόεδρος. Και τώρα έχει το λόγο κυρία Κλειβέτη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Κάσα, ε, που συνεργαστήκαμε πάρα πολύ παραγωγικά για αυτή την έκθεση. Πολύ σημαντική η έκθεση αυτή και συμπληρώνει κάποιες αποφάσεις που ήδη έχουμε λάβει εδώ στο Κοινοβούλιο και αναφέρομαι ε, στην απόφαση σε σχέση με το Erasmus, ΣΥΝ. δηλαδή ε, για την απασχολή των νέων και την πράσινη οικονομία σε σχέση επίσης και με τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν ε, όσον αφορά τις πολιτικές που θέλουμε να ε, ασκήσουμε όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Από σήμερα μέχρι το 2030 θέλουμε να αρχίσουν να τρέχουν διάφορα προγράμματα, θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα, γιατί πολλές ευκαιρίες προσφέρονται σε ένα ζήτημα τόσο σημαντικό για όλο τον κόσμο. τίτλοι σπουδών και λοιπά, όλα αυτά θα πρέπει να καλυφθούν. Τροπολογίες, ε, έχουμε πολλές με τις οποίες συμφωνούμε, οπότε και θα υπερψηφίσουμε την έκθεση. Λάμπερτ, ευχαριστώ. Όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες, έχουμε πέντε στις οποίες καταλήξαμε. are now moving in as compared to the, the original from the rapport. Έτσι, στην ε, συμβαστική D. 4. Συμβαστική 4 ή τη D, εκεί έχουμε την αρχική πρόταση, η οποία αφορούσε το πώς θα γίνει η ε, αλλαγή από την αρχική ε, ιδέα σε σχέση με αυτή την πράσινη οικονομία, γιατί μιλάμε για κάποιους ε, τομείς ενεργειακής έντασης και να δούμε πώς θα προσαρμοστούν ε, στις ε, διαφορετικές συνθήκες οι εργαζόμενοι. Να δούμε πώς εδώ θα προστατεύσουμε τις θέσεις απασχόλησης αλλάζοντας κάποιες ευρύτερες πολιτικές όσον αφορά με τις ε, ποσοστώσεις όσον αφορά τις ε, βλαπτερικές εκπομπές και την ε, ενεργειακή πολιτική. Στο Ι e έχουμε εδώ μια διάταξη συμβαστική πάρα πολύ δύσκολη. Συμβαστική τροπολογία, συν τροπολογία συγχωνεύτηκαν εδώ. Και εδώ ασχολούμεθα με τις ε, με τους τομείς εκείνους της βιομηχανίας που έχουν να κάνουν με ένταση ενεργειακή, την ενεργειακή πολιτική που ισχύει. Οπότε για το D και το E έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, ε, οι άλλες μας ικανοποιούν, ε, κατανοούμε ότι έχει καταβάλει προσπάθεια ο εισηγητής. γιατί έπρεπε να εξετάσει το τι θέλει η δική του πολιτική ομάδα και οι άλλε πολιτικέ ομάδε. Οπότε σα για τι επιφυλάξει μα, γι' αυτό και δεν έχουμε προσυπογράψει ω ομάδα αυτέ τι ε, τροπολογίε. Σα ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστώ του συζητητέ, του συναντέλφου, ε, του και του συζητητέ. Ε, εστιάσαμε την προσοχή μα στο καθήκον μα. Δηλαδή, το καθήκον μα είναι σε αυτό το τόσο σημαντικό έγγραφο για την ενέργεια και το κλίμα, να εστιάσουμε την πολιτική μας και στην κοινωνική πολιτική. Και Επίσης ε, να δούμε κατά πόσο υπάρχει ένας κλιματιστόχος, δύο, τρεις ή και περισσότεροι ακόμα. Ευχαριστώ όλους ε, θερμά γιατί αυτά ήταν πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι επιτύχαμε καλές συμβαστικές ε, προτάσεις και αυτά όλα δείχνουν ότι δεν δίστανται τόσο πολύ οι απόψεις μας όταν πρόκειται για τα κοινωνικοπολιτικά θέματα. Επόμενη στόχη στην ε, κλιματική αλλαγή είναι σημαντικό να οριστούν ε, μέχρι το 2030. Οι συμβαστικές προτάσεις είναι μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στον τομέα για την πράσινη τεχνολογία αφενός και αφετέρου ε, στον κίνδυνο ε, που είναι πολύ σημαντικός για τους απασχολούμενους να μην υπάρχουν στόχοι που είναι ανέφικτοι και που σε τελική ανάλυση στοιχίζουν θέσεις απασχόλησης. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να είναι στόχος της Επιτροπής. Γι' αυτό λοιπόν ε, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το ότι καταλήξαμε σε καλές συμβαστικές προτάσεις και σε μια πολύ καλή εισήγηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Ο εισηγητής μας. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Κατανοώ τη θέση της κυρίας Λάμπερτς, αλλά ξέρετε ότι δεν μπορούν όλοι να είναι ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε λύση και αν προκρίνουμε. Θα τα καταφέρουμε καλύτερα την επόμενη φορά. Πρόεδρος. Ε, ναι, αλλά άμα η επόμενη φορά είναι για το, το 2040... Ε. Τέλος πάντων. Σταματάμε εδώ. Για το σημείο 8 Θα σας παρουσιάσω το σχέδιο επιστολής που απευθύνουμε στο πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για την προσαρμογή ε, των άρθρων 90 ε, ε, και 92 της συνθήκης για μια σειρά νομικών πράξεων για την προσφυγή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για το Omnibus 3. το Συζητήσαμε σε προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας αυτό το ζήτημα και με τη γραπτή διαδικασία καταφέραμε να συμφωνήσουμε για την έγκριση μιας πολύ σημαντικής τροπολογίας. Ε, ο Τσάμπα Όρη ε, ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την τροπολογία διότι ανησυχούσε ε, για την ε, προθεσμία μέσα στην οποία έπρεπε να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αιτήματά της για την ευθυγράμμιση με αυτά τα άρθρα της συνθήκης. Οι πράξεις ε, κατά εξουσιοδότηση φτάνουν πάντοτε στο τέλος της θητείας με κάποιο τρόπο. Εδώ πρόκειται για την ευθυγράμμιση τριών νομικών πράξεων που ε, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της δικής μας ε, Επιτροπής, ε, αλλά δεν μας ζητήθηκε γνωμοδότηση. Και κατά την εξέταση του Omnibus 1, συνειδητοποιήσαμε πως έλειπε η δική μας γνωμοδότηση. από απουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μπορώ να σας πω ότι συμφώνησαν όλοι οι συντονιστές να στείλουμε αυτή την επιστολή στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την ενσωματώση στις δικές της εργασίας. Ε, για, στο πρώτο παράρτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ευθυγράμμιση των μέτρων μέσω ε, πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Στο παράρτημα 2 προτείνει ευθυγράμμιση των μέτρων πρακ με εκτελεστικές πράξεις και επί τη βάση της έκθεσης Τσάγερ που εγκρίθηκε ε, ήδη από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θεωρούμε ότι τα μέτρα ΠΡΑΚ θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται μέσω πράξεων ε, κατά εξουσιοδότηση και όχι εκτελεστικών πράξεων. Οπότε προτείνουμε ε, να καταργηθεί η πρόταση για το παράρτημα 2 και αυτά τα μέτρα να ενσωματωθούν στο παράρτημα 1 ώστε να υπαχθούν στο καθεστώς ευθυγράμμισης μέσω πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Αν παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υιοθετήσει πιο ευέλικτη προσέγγιση ε, και δεδομένου του εξαιρετικά τεχνικού χαρακτήρα των σημείων εφόσον πρόκειται για τις ε, ημερομηνίες διαβίβασης ε, των πληροφοριών και το μορφότυπο διαβίβασής τους θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη θέση μας όπως θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. δεν μπορούμε να υπερβούμε την πενταετία για τις πράξεις κατεξουσιοδότησης σε καμία περίπτωση και... Ε, θέλουμε να αναφέρουμε στον κύριο Όρη ότι πρέπει να αποφύγουμε την επικάλυψη αυτών των εξελίξεων με την προεκλογική εκστρατεία ή τις ευρωπαϊκές εκλογές ή την ε, δημιουργία των νέων επιτροπών. Η διαδικασία θα είναι διαφορετική ανάλογα με την ε, κάθε επιτροπή. Ε, την αρμόδια επιτροπή, οπότε ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητείτε γνωμοδότηση από την επιτροπή μας για ε, οποιαδήποτε τέτοια ευθυγράμμιση. Υπάρχουν σχόλια? Όχι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Είναι διαδικαστικό το ζήτημα. Σημείο 9. Θα στείλουμε την επιστολή, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 9. Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Μεταφορών πρόταση ε, κανονισμού ε, κανονισμός 718 του 1999 για τους κανόνες ναυσιπλοείας για τις εσωτερικές ε, πλωτές ε, οδούς η Γιούτα Στάινρουκ είναι η συγγήτριά μας. Ε, θα της δώσω το λόγο ε, για την εξέταση ε, του σχεδίου γνωμοδότησης. Παρακαλώ. Äh, Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής. Ε, για αυτή την πρόταση συζήτησα τόσο με τα συνδικάτα όσο και με τα ε, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ναυσιπλοείας. 35 ε, εκατομμύρια ευρώ ε, πρέπει να είναι το απόθεμα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό από το 1989 όμως δεν ισχύει. Η δική μου λοιπόν η πρόταση λέει ότι θα πρέπει να αναδιατυπωθεί το κείμενο, να έχουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες οι οποίοι θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο αυτό και στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού των στόλων ε, πρέπει να βελτιωθεί οπωσδήποτε η επαγγελματική κατάσταση των απασχολούμενων. Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να υπάρχει και η δυνατότητα ε, πρόορης συνταξιοδότησης. Το τρίτο σημείο αφορά στον τεχνικό εξυγχρονισμό ε, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, αυτό στο μέλλον θα είναι ε, υποχρεωτικό και το Ταμείο θα προβλέπει ε, και σχετικά προσόντα για τα μέλη των, ε, για το πλήρωμα των σκαφών. Κατόπιν γίνεται λόγος και για διάφορες αλλαγές μπορούν να γίνουν σε ένα σκάφος, αυτές όμως πρέπει να κοινοποιούνται. Και εγώ παραθέτω ότι οι πληροφορίες, ε, κυρίως ε, για την πρόορη συνταξιδότηση και τη μερική απασχόληση, πρέπει να προωθηθούν. Αυτό πολύ συγκεκριμένα σημαίνει ότι τα συνδικάτα ε, θα πρέπει να μπορούν να οργανώνουν ενημαρωτικές εκστρατείες από κοινού με τα ταμεία τα αρμόδια Σημαντική προϋπόθεση είναι τα κονδύλια να χορηγούνται προς όφελος των απασχολούμενων και των επιχειρηματιών. Για μένα λοιπόν εδώ είναι απολύτως απαραίτητο να συμμετέχουν επίσημα οι κοινωνικοί εταίροι στην χορήγηση των κονδυλίων. Γιατί οι κοινωνικοί εταίροι τόσο επιχειρήσεις όσο και τα συνδικάτα γνωρίζουν τα προβλήματα. Ως εκ τούτου εγώ έχω προτείνει τις εξής ε, τροπολογίες. Στο άρθρο υπαριθμών 1 επιθυμώ ε, τα κράτη-μέλη από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους να μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα κοινωνικά μέτρα. Στο πρώτο εδάφιο λέω ότι θα πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών και μέσα από ε, εκ νέου κατάρτιση ή ε, πρόορη συνταξιοδότηση. Στο δεύτερο εδάφιο θέλω να καταστήσω σαφές ε, όλα αυτά να υπάρχουν και για τα πληρώματα των πλοίων. Δηλαδή ε, όχι μόνο η δυνατότητα περαιτέρω κατάρτισης, αλλά και πρόορη συνταξιοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη προβλέπει κάτι τέτοιο για τις επιχειρήσεις. Στο τρίτο εδάφιο θέλω να καταστήσω σαφές ότι όλα τα μέλη ε, του πληρώματος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καλύτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στο τέταρτο εδάφιο ε, το διόμορφοι, ε, θα πρέπει να το αντικαταστήσουμε, να αντικαταστήσουμε τη λέξη αυτή αυτή ε, με σκάφη και μεγαλύτερου μεγέθους. Ε, τους κοινωνικούς εταίρους τους αναφέρω σκόπιμα διότι η αρχική έννοια οργανώσεις για μένα ήταν ε, πάρα πολύ γενική. Κοινωνική εταίρη σημαίνει και αναγνωρισμένες ε, επαγγελματικές ενώσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη εμπειρία στην εκπροσώπηση των συμφερόντων. Στο πέμπτο εδάφιο γίνεται λόγος για τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας που πρέπει αυτή να συμβαδίζει με τη βελτίωση των, ε, της προστασίας από ατυχήματα, από επαγγελματικά ατυχήματα. Αυτό μπορεί να το εννοεί η Κομισιόν, αλλά δεν το έχει καταγράψει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ επιθυμώ να υπάρχει σαφής ε, διατύπωση. Αυτές είναι οι προτάσεις μας και χαίρομαι, οι προτάσεις μου και χαίρομαι πάρα πολύ για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ο κύριος Φίλιπ ε, Ντεπάκα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ την είπε και για την ε, δουλειά του. Από ό,τι φαίνεται ήταν αξιόλογη η πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέρασαν κάποια δύσκολα χρόνια και ακόμα υπάρχουν προβλήματα, οπότε και γι' αυτό και θα πρέπει επιτέλους κάτι να κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε το βάρος στην καινοτομία ε, στο πώς ε, τα, τα σκάφη θα είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. Είναι, είναι πολύ αξιόλογη τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. των σκαφών. Αυτό προτείνεται. Να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογική πρόοδο. Πρεκοδότηση δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, οπότε θα πρέπει να είναι καλά στοχευμένες οι οι ενεργειές μας ε, άρα πρέπει να προσπαθήσουμε προσεκ... Ε, πολύ συγκεκριμένα να μην έχουμε δέκα προτεραιότητες ας πούμε να προσέξουμε τα πιο ε, σημαντικά θα πρέπει οι πόροι να πάνε στα πιο σημαντικά και καινοτομία, εξυγχρονισμός, στόχευση ενημέρωση ο πλευρά τεχνολογία και επικαιροποίηση, οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στην εκπαιδεύση του θέματο, γιατί ο χρόνο ε, πιέζει και ελπίζω να κλείσει το θέμα, να συμφωνήσουμε τέλο πάντων σε πρώτη ανάγνωση πριν το τέλο τη ε, ε, θητεία. Άρα, καλά στοχευμένε ενέργειε και το συντομότερο δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε για την εσωτερική ναυσιπλοεία τους πόρους που υπάρχουν. Θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει πρόεδρος. Όχι. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Σύγεται, έχει πάλι το λόγο. Θα ήθελα ε, σύντομα να επισημάνω κάτι στον κύριο Ντεμπάκαρτ. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα ε, δεν έγινε απορρόφηση των κονδυλίων. Από το 99 πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε έτσι ώστε στο πλαίσιο των στόχων του προγράμματος να περιζόμαστε στην εσωτερική ναυσιπλοεία, να προσπαθούμε να ρυθμίσουμε την αγορά και όλα αυτά να γίνονται με, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να απορροφώνται τα κονδύλια. Αυτός πρέπει να είναι στόχος μας. Μέχρι τώρα ε, τα κονδύλια, επειδή ε, ήταν ασαφής η κατάσταση, όπως σας είπα δεν ανακλήθηκαν και αυτό είναι το κύριο μέλημα του κανονισμού. Πολύ ωραία. Οπότε, αρχίζει η προθεσμία υποβολή των τροπολογιών για το σχεδικημένο σας Έχουμε ήδη 8 τροπολογίες και η προθεσμία θα είναι 7 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Αυτές οι τροπολογίες θα συζητηθούν 22 και 23 Ιανουαρίου και θα ψηφίζουμε 12 και 13 Φεβρουαρίου. η Επιτροπή Μεταφορών παράλληλα θα κινηθεί και θα ψηφίσει 20 Φεβρουαρίου. Και το ζήτημα θα κατέβει στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Τελειώσαμε αυτό το σημείο της ημερικής διατάξεως. Και πάμε τώρα στο 10. Θα πρέπει εδώ πέρα να σα παρουσιάσω τι κρατήρε γραμμέ για τι πολιτικέ απασχόλησεις των κρατών μελών. Ρίξτε μια ματιά στο κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που από αυτό το Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ σύντομο γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια τυπική διαδικασία. χρειάζονται τη σχετική προσαρμογή. Στην αρχή της θητείας μας εγκρίθηκαν αυτές οι συνθήσεις γραμμές, αλλά κάθε χρόνο πρέπει να επεξεργαζόμαστε τις ε, ειδικότερες διατάξεις στις 11 Ενάτου οι συντονιστές αποφάσισαν να εφαρμοστεί η απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση του κειμένου. Σύμφωνα με το άρθρο 46, παραγωγός 1 του κανονισμού λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Οπότε για μια πρώτη συζήτηση μας προσφέρει τη δυνατότητα να ελέγξουμε το κείμενο χωρίς τροπολογία. Σας διαβάζω το άλλο αντίκτυπο του κανονισμού. Στα αγγλικά. Δείτε στα αγγλικά έχω το κείμενο. Λέει το τέξι, ένα τέξις. Εάν δεν ενίσταται ένας τουλάχιστον βουλευτής μπορεί ο Πρόεδρος να υποβάλει προς έγκριση το σχέδιο κειμένου την πρόταση. Στην περίπτωσή μας αυτό θα πρέπει να γίνει τον Φεβρουάριο. Οπότε θα πρέπει να συμφωνήσει το 10% δηλαδή 5 τακτικά μας μέλη. Οπότε μπορούμε ίσως να ανοίξουμε μια προθεσμία για τροπολογίες 14 πρώτου το μεσημέρι. Από τότε είχαν αρχίσει να υποβάλλονται και θα συζητηθούν αυτές το 22 Ιανουαρίου του 2014. Η δε έκθεση θα ψηφιστεί όταν συνεδριάσει η Επιτροπή μας στις 23 Ιανουαρίου. Αν όμως δεν υποβληθούν τροπολογίες θα θεωρηθεί ότι το κείμενο εγκρίνεται. Σας υπενθυμίζω το ιστορικό πλαίσιο πρόκειται για εφαρμογή του άρθρου 148 παράγραφος 2 της ε, συνθήκης το οποίο προβλέπει την ε, έγκριση αυτών των κατευθυντηριογραμμών. Si, s'il n'y a pas d'objection Je vous propose de ne même pas ouvrir la procédure de délai. Αν επομένως δεν υπάρχει κάποια ένσταση, να μην ανοίξουμε καν προθεσμία έγκρισης τροπολογιών και να προχωρήσουμε έτσι ευθύ αμέσω. Έχει κάποιος κάποια ένσταση, θέλει κανείς τον λόγο, όχι. Γιατί το συγγραφεί κάτι αφού πρόκειται την απασχόληση. Τι σχέση έχουν αυτές οι διαδικασίες με την πραγματικότητα, αφού ξέρουμε πώς έχει κατάσταση σε όλες τις χώρες. Ε, ευχαριστώ. Οπότε τελειώσαμε το σημείο 10. Έχει κάποιος κάτι για τα διάφορα. Έχετε δύο λεπτά για να το προτείνετε. Bien. Euh, les deux minutes... Καλώς. Υπολογίζω πέρασε το δίλεπτο. Οπότε τώρα αρχίζουν οι ψηφοφορίες. Προς υπόμνηση. Επειδή στο 10 δεν υπήρχε κάποια αντίρρηση, θεωρούμε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών εγκρίνονται. Σήμερα με το άρθρο 46 παραγραφός 1 του κανονισμού. 11. Έχετε όλη την κάρτα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πάμε στο σημείο 11. ολοκλήρωση, επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αρρωγής προς τους απόρους. Είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει για μία δήλωση στην Ολομέλεια μία εξήγηση για τα κοινωνικά παντοπολία Κατά τη γνώμη μου όμως ε, γεννά πολλά ερωτηματικά ε, προς το παρόν τουλάχιστον η δήλωση του Επιτρόπου. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι την Ολομέλεια. Θα δούμε πώς θα απαντήσει ο Επίτροπος στην Ολομέλεια. Εάν ε, δεν ζητάει κανείς το λόγο, προτείνω να ψηφίσουμε το σύνολο της έκβασης των διαπραγματεύσεων. Παρακαλώ, άρχιε την ψηφοφορία. Better and better again. Marianne Harkin, if you want to vote, you better be... Marianne Harkin, αν θέλεις να ψηφίσεις γρήγορα. But otherwise I can close the vote. Ότι θέλω να κλείσω, κλείσω το, την ψηφοφορία τώρα γρήγορα. Ορίστε. Κύριος Πυρμανιάς. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Δεν περιμένω άλλο. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 32 ψήφισαν, 30 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια προς την κυρία Κοστέλο και ολόκληρη την ε, ομάδα ε, που ασχολήθηκε με τις διαπραγματεύσεις. Σημείο 12 είναι η επιστολή που σας παρουσίασα νωρίτερα. Επιστολή προς ε, την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για το Omnibus 3 για την προσαρμογή στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο. Προτείνω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ, αρχής ψηφοφορία. Πέρας. 34 ψήφισαν, 31 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. 13 τώρα. Ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ε, προ την Επιτροπή ΙΜΚΟ που συνέταξε ο Μάρτιν Κάσλερ για το πρόγραμμα Solvit. Ε, συμβαστική 1 για την πρώτη παράγραφο. Πέντε πολιτικών ομάδων. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 1, συμβαστική Β των 5 ιδίων πολιτικών ομάδων υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Παράγραφος 2, συμβαστική Γ, οι 5 πολιτικές ομάδες υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Παράγραφος 3, συμβαστική Δ των 5 ιδίων ομάδων υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 13 τώρα της Αντιγόνης Παπαδοπούλου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα χωρίς το encourages member states to strengthen synergies between Solvit and the respective administration for the better coordination of social security systems. Χωρίς αυτά, αυτή την αράδα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα, για την προσθήκη αυτής αράδας, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 4, συμβαστική ε, 5 ομάδων υπερκατά. εγκρίνεται. Μετά, παράγραφος 4, συμβαστική J, υπέρ αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5, συμβαστική F, 5 ομάδες υπέρ εγκρίνεται. Μετά, συμβαστική G από τις 5 ίδιες ομάδες υπερκατά. εγκρίνεται. Παράγραφος 6, συμβαστική H των ίδιων ομάδων, ε, πολύ ωραία συνεργασία τους υπέρ κατά αποχές. Ε, γκρίνεται, συμβαστική I, πάλι της ομάδας υπέρ κατά Ε, γκρίνεται. Τελειώσαμε με την ψηφοφορία για τις τροπολογίες. Ψηφίσουμε το σύνολο της νομοδότησης με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχη ψηφοφορία. Πέρας. 35 ψήφισαν, 35 υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια, κύριε Κάσλε. Σημείο 15 τώρα. Σχέδιο γνωμοδότησης σε Μεταφορών για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. Πρόκειται για σχέδιο γνωμοδότηση του κυρίου Τεμπάκερ. Ψηφίζουμε όχι για το σχέδιο γνωμοδότησης, εγώ νομίζω, αλλά για το σχέδιο κανονισμού. προτείνεται απόρριψη του σχεδίου κανονισμού που έχει συνταχθεί υπό τη μορφή τροπολογίας παριθμών 6 τη κυρία Σρέντερ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Tout le monde Ψήφισαν όλοι πέρας. 18 υπέρ, 18 κατά. Μία αποχή. Narrow escape το λέμε αυτό αγγλιστή. Φτηνά τη ε, ισοψηφία και απορρίπτεται. Πολύ χαίρεται ο συγητής. Παράγραφος 2, σημείο Γ, τροπολογία 27, Richard Howitt. Τροπολογία για την κατάργηση τμήματος υπέρ κατά αποχές παλήθευση εφόσον είχαμε το προηγούμενο αποτέλεσμα. Ψήφιστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας. 19 υπέρ, 18 κατά. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Το άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο Γ καταργείται. Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο Δ. Τροπολογία 28, Ρίτσαρτ Χάουιτ, επίσης ε, ζητείται κατάργηση του σημείου, διαγραφή του σημείου. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Πέρας. 19 υπέρ. 18 κατά καμία αποχή. Διαγράφετε το δέλτα εδάφιο. Ε, στο G, ε, σημείο G, ε, τροπολογία 29, Χάουιτ και 30 της Στάινρουκ, ε, ταυτόσημες ε, και ο στόχος είναι η διαγραφή του σημείου. με ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Παρακαλώ. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Πέρας. Εγκρίνεται 19 ψηφί υπέρ 18 κατά και καμία αποχή. Σημείο H. Τροπολογία 31. it. Ο στόχος είναι η διαγραφή του σημείου H. Παρακαλώ με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 19 pour, 18 contre, 0. 19 ε, υπέρ 18 κατά, καμία αποχή, διαγράφεται το σημείο H. 2-1, ε, εδάφιο 18α, τροπολογία 32, Ζαμπιέ είναι κατά, ο εισηγητής, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία και άρα η πρώτη παράγραφος τροποποιείται αντιστοιχώς σημείο 2, ε, τροπολογή 33 Χάουιτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, τώρα άρθρο 2 παράγραφος 1 ε, σημείο 18α Jean Pierre 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Άρθρο 2, παράγραφος 1, μετά το 18, τροπολογία 35, Ρίτσαρτ Χάουιντ υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 4, παράγραφος 1, τροπολογία 36, Γιούτα Στάινεροκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4-2 ε, στην εισαγωγή, τροπολογία 37, Ελίζα Schroeder υπέρ, κατά αποχές παλήθευση, παρακαλώ, για την 37. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Πέρας. 19 ψήφοι υπέρ 18 κατά καμία αποχή. Την πλειοψηφία με τον αριθμό των μελών που έχουμε. Άρθρο 4, παράγραφο 2, σημείο α, τροπολογία 38. Σρέντερ είναι υπέρ ο εισηγητής, υπέρ κατά αποήχε εγκρίνεται. 4-2 εδάφιο γάμα, τροπολογία 39, σρέντερ, είναι υπερουσίγητης υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται, τροπολογία 40, Ζος Μπάχ, είναι συμβατή, η τροπολογία την ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται, άρθρο 4 παράγραφος 2, μετά το σημείο Δέλτα, τροπολογία DA, ε, τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ κατά εγκρίνεται, άρθρο 4 παράγραφος 3, τροπολογία 44. Σέρτζιο Παόλο και Φρανσέσκο Σιλβέστης. Υπέρ κατά αποχές ε, επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 20 ψήφοι υπέρ 16 κατά, όντω εγκρίθηκε. Άρθρο 5, παράγραφο 2. Μετά την υποπάραγραφο 2 έχουμε την τροπολογία 45 στρέντερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 6, παράγραφος 1, μετά το σημείο Β, τροπολογία 46, Ρίτσαρτ Χάιουντ υπέρ κατά εγκρίνεται. Άρθρο 7, παράγραφος 2, τροπολογία 47, δεν γίνεται παραδεκτή, ούτε και 48, ούτε και 49, ούτε και 50, ούτε και 51. 52 τώρα για την 8, 1, α, Σρέντερ, είναι υπέρ, ο υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 8, παράγραφος 1, μετά το σημείο Γ, τροπολογία 53, Χάουιτ υπέρ, κατά απόχέ. εγκρίνεται. Άρθρο, έτροπολογία ε, τροπολογία 54 δεν είναι παραδεκτή και πάμε στο άρθρο 8, παραγραφό 6, τροπολογία 55, Χάουιτ, προτείνει η διαγραφή του σημείου υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. κατόπιν έχει υποβληθεί... Εντάξει, ωραία, θα το ελέγξω, θα σας πω γιατί έχω δίκιο, γιατί ξέρω ότι έχω δίκιο. Ξέρω, ξέρω γιατί το ζητάτε για τις διαπραγματεύσεις. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 14 ψήφοι υπέρ, 23 κατά, μία αποχή. Όπως το αναμέναμε, δεν εγκρίνεται η τροπολογία. Ah euh, την προφορική τροπολογία δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε δεν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε αν είχε εγκριθεί 55. Εφόσον όμως ε, δεν εγκρίθηκε μπορούμε να την ψηφίσουμε. Υπάρχει... Θέλετε να τοποθετηθείτε για την προφορική τροπολογία του κυρίου Χάουιτ. Όχι. Ωραία θα την ψηφίσουμε. Παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Θέλετε παλήθευση κύριε Χάουιτ. Έτσι το βλέπω εγώ. Έτσι που σας κοιτάζω, πολύ ωραία. Επαλήθευση, παρακαλώ. Πέρας. 31 υπέρ 7 κατά καμία αποχή ξεκάθαρα εγκρίνεται η προφορική τροπολογία. Αντίθετα, η 56 του George Bach καταπίπτει ως εκ τούτου. Και άρα φτάνουμε στο άρθρο 10 παράγραφος πρώτη συμβαστική ε 4 πολιτικών ομάδων κατα αποχές. Εγκρίνεται. Ε, άρθρο 10 παράγραφος 2 συμβαστική ε α τριών ομάδων υπερκατά αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 10 παράγραφος 3. 64 της κυρίας Στάινερο και υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 Χάουιτ, παρακαλώ υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Να το άρθρο 1066 Steiner υπέρ κατά αποχές. Επαλήθευση για την τροπολογία 66 ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. 19 προς 19 απορρίπτεται. Άρθρο 11, η 67 του κυρίου Χάουιτ, υπέρ. Κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται κεφάλαιο 2α νέο, τροπολογία 68 Ρίτσαρτ Χάουιτ, είναι κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Ε, άρθρο 12, παράγραφο 3, τροπολογία 69, Ζαν υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 12. Μετά την παράγραφο 7, τροπολογία 70, ε, οντί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, άρθρο 15, παράγραφος 1, η 71, Σρέντερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο... Α, εντάξει, και okay, επαλήθευση για την 71. De tous les votes. Ήρθε η ώρα για τα χριστουγεννιάτικα δώρα και με ζητάτε επαλήθευση για όλες τις τροπολογίες. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 19 προς 19. Καλά κάνατε και ζητήσατε επαλήθευση, αλλά εγώ καλά έκανα που σας έλεγα εξ αρχής ότι απορρίπτεται. Λοιπόν, για το εισαγωγικό τμήμα του άρθρου 16, τέσσερις πολιτικές ομάδες συμβαστικές υπέρ. Χειρότερα θα ήτανε απαντώντας λέει η Πρόεδρος σε κάτι που δεν άκουσαν οι διερμηνείς. Συμβαστική F, τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, άρθρο 16, παράγραφος 1, μετά το σημείο Γ, 75 στα και υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Εντάξει, ε, εάν το ζητήσει η συντάκτηρια της τροπολογίας, εγώ με τα χαράς να κάνω την επαλήθευση. Παρακαλώ λοιπόν, για την 75... Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Μένα μου φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο πως εγκρίνεται. 32 είναι οι ψήφοι υπέρ, 7 κατά, καμία αποχή. Άλλαξαν τα πράγματα, καλά κάναμε και παληθεύσαμε διότι εγκρίνεται. 76 Τζος Μπαχ, άρθρο 16 υπέρ κατά αποχές, ε, ξεκάθαρα εγκρίνεται. Άρθρο 17, τροπολογία 77, ε, δεν είναι παραδεκτή, το ίδιο και η προφορική τροπολογία, το ίδιο και 78, 79 και 80. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις, 5, τροπολογία 1, το εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 το εισηγητή μετά το εκτιμώντας 5 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την τροπολογία 2 άρχιδη ψηφοφορία. Ψήφισαν άλλοι 21 υπέρ 18 κατά καμία αποχή. Εγκρίνεται. Ε, το ιδεολογική σκέψη 6 ή 7 του κ. Χάβιτ υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται ε, τιολογική 7 συμβαστική α 4 ομάδων υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στην τροπολογία 10 μετά την αιτιολογική 7. Χάουιτ υπέρ κατά αποχές ε, ε, επαλήθευση. Εντάξει. Για την τροπολογία 10. Επαλήθευση παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας. 24 υπέρ, 15 ε, κατά καμία αποχή, ξεκάθαρα εγκρίνεται. Ε, μετά το, την αιτιολογική 9, η τροπολογία 11 του Χάιουιτ επίση υπέρ, ε, κατά αποχές, απορρίπτεται. Καταπίπτει η 12 και φτάνουμε στην αιτιολογική 14, συμβαστική β, 4 ομάδων υπέρ, κατά αποχές Εγκρίνεται αιτιολογική 19, συμβαστική ΣΥΔΙ, τριών ομάδων υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται αιτιολογική 19, ζώος Μπαχ 19 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται, η 20 δεν είναι παραδεκτή. Και μετά την αιτιολογική 20 ψηφίζουμε την 21 Χάουιτ υπέρ κατά αποχές. Υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Χάουιτ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 δεν είναι παραδεκτή και άρα συμβαστική δέλτα μετά την αιτιολογική 31, τέσσερις πολιτικές ομάδες υπερκαταποχές εγκρίνεται μετά την αιτιολογική 31 η 26 δεν είναι παραδεκτή ψηφίζουμε το σύνολο της μαμοδότησης. ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ ψήφισαν όλοι πέρασε 25 υπέρ, 14 κατά καμία αποχή. Εντάξει, δεν πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένο ο εισηγητή κατά το ίμιση. Συγχαρητήρια παρόλα αυτά. Σημείο 16. Θα ψηφίσουμε τώρα την ε, έκθεση που αφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος και την Επιτροπή Ήτρα κυρίως αρμόδιες επιτροπές και αφορούν αυτό το πρόγραμμα της πολιτικής. Sur un rapport d'initiative s'agissant du cadre pour euh, les politiques en matière είναι το πλαίσιο για τις πολιτικές του κλίματος και ενεργείας. Με ορίζοντα το έτος 2030 η 1 από τέσσερις πολιτικές ομάδες σχετική συμβαστική που ονομάζεται Α. Ε, Α1, ε, τροπολογία 3, Κρίστενσεν εγκρίνεται, τροπολογία 4, Κλιβέτη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 5, Κρόιτσμαν, υπέρ κατά ε, αποχές, ποιοι είναι υπέρ Αληθεύει η Πρόεδρος. Είναι κατά αποχές. Την παρέλευση για το 5. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 21 ψήφι υπέρ, 17 κατά και μία αποχή εγκρίνεται. Ε, 6 εγκρίνεται. 7 κλειβέτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 κλειβέτη. Με προφορική τροπολογία δεν έχετε καμία ένσταση και επομένως ε, πάμε στο 8 υπέρ κατά αποχές. Επαλήθευση, γιατί δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, δεν βγαίνει ψήφι. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1. Δέλτα. 9. Κλειβέτη υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Συμβαστική Β. Από τέσσερις πολιτικές ομάδες υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Μετά έχουμε την παράγραφο 2. Τροπολογία 12. Κρίστανσεν, Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Συμβαστική Γ. Από τέσσερις πολιτικές ομάδες υπέρ κατά αποχές. 3. 16. Κρόιτσμαν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Συμβαστική δέλτα. Τρεις πολιτικές ομάδες υπέρ κατά εγκρίνεται. 19. Κλειβέτη. Σε διερμήματα αιτήσει του ΕΛΚ. Μέχρι εκεί που λέει ε, incentive sector στον ελληνικό κείμενο Απορρίπτεται. Ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα της 19. 20 απαράδειγμα Δεν την ψηφίζουμε. 5. Παράγραφος 5. Συμβαστική ε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατόπιν το 25 κλειβέται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του κειμένου. Ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίζουμε τώρα. Ψηφίσανε όλοι. Πέρας. 39 υπέρ. Ουδής κατά. Αποχές. Συγχαρητήρια προς ε, τον εισηγητή ή μάλλον την, τον εισηγητή, τον κύριο Κάσα. Τώρα, η επόμενη ψηφοφορία. Η τελευταία για σήμερα. Αφορά το σημείο 17. dont nous sommes convenus en réunion des coordinateurs et sur nous avons euh, pu... Euh, έχουμε αυτές τις τροπολογίες ε, που προήγησαν τη συνάντηση των ε, ε, συντονιστών και έχουμε τώρα αυτή την έκθεση που αφορά την ισότητα ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι έκθεση του 2012. qui seront déposées en notre nom euh, directement au sein de la commission. sur le paragraphe un nous sommes. Πρώτη παράγραφος. Τροπολογία 3 κλειβέτη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5. Κλειβέτη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 οι φιλελεύθεροι έχουν ζητήσει κατά διέρεση ψηφοφορία. Το πρώτο, μέχρι εκεί που λέει developments. Υπέρ κατά απορρίπτεται το επόμενο, το υπόλοιπο κείμενο υπέρ κατά εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 7. Μπαλτατσίνο. Υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 8, κλειβέτη. Σε δύο τμήματα, το πρώτο αιτήσει των φιλελευθέρων. Κατά τη ψηφοφορία υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχέ. Το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Στη συνέχεια μετά την τέταρτη παράγραφο έχουμε την τροπολογία 9. Υπέρ κατά, τι είναι κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 10. Θα κάνουμε όμως πρώτα επαλήθευση για το 9. Ψηφίζουμε σύφισεν όλοι πέρας 15 19 4 αποχήσ απόλυτοι 10 κλιβέτηι πέρ κατά αποχήσ ηγρίντε 11 κλιβέτηι πέρ κατά αποχήσ ηγρίντε 12 κλιβέτηι πέρ κατά αποχήσ ηγρίντε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 κλειβέτη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 κλειβέτη σε δύο τμήματα. Όπως ζήτησε το ΕΛΚ. Και ψηφίζουμε το σύνολο του 15. Χωρίς τη φράση Α, όχι, όχι, λέει η Πρόεδρος. Έχουμε επομένω δύο τμήματα και το πρώτο τμήμα θα είναι χωρίς τη φράση που λέει θα αναγνωρίζει την προσθέμενη αξία των γυναικών ή στον χώρο εργασίας. και έχουμε επίση και προφορική τροπολογία του ΕΛΤ. Άρα, πάμε στο πρώτο τμήμα του 15 όπω τρόπο. Πλημπολογική τροποποιήθηκε. Την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Είναι υπέρ τη προσθήκη των λέξεων που είπαμε ότι θα προβλέπονται. Απορρίπτω και αυτή η πρόταση τώρα. Τροπολογία 16 Μπαλτατσίνο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 17 της ε, Βαλτατσίνου υπέρ 18 της Ιδίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 Βαλτατσίνου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Παραγραφός 10, τροπολογία 20. Μπαλτατσίνου. Εγκρίνεται. Όσον αφορά την αιτιολογική σε γάμα, υπαριθμών 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κατόπιν η αιτιολογική F, η τροπολογία 2, υπέρ κατά Και με αυτές τις τροπολογίες ολοκληρώσαμε τις ε, ψηφοφορίες και πάμε στο σημείο 19. Sur notre rapport d'initiative. Έχουμε την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που αφορά τον ρόλο και τις δραστηριότητες της Τρόικα. FMI dans les pays du programme de la zone euro. Euh, il s'agit d'un rapport... Πρόκειται για κάποια έκθεση την οποία έλαβε ως εισηγητής ο Αλεχάνδρο Θέργας. Είπαμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει μια έκθεση που αφορά το ίδιο ζήτημα. Αλλά η διάσκεψη των πρόεδρων στις 12, του δεν συμφώνησε. Deux commissions associées. En revanche, elle nous euh, Και αντί να γίνει από κοινού και εκ παραλλήλου, θα γίνει τελικά, θα γραφτεύσει κάθε συναρμόδια επιτροπή χωριστά. Και έτσι ανέλαβαμε αυτή την έκθεση τη πρωτοβουλία και τώρα σκητάλη στον εισηγητή. Como usted ha dicho, tenemos la oportunidad de hacer informe de iniciativa, pero en la reunión de esta mañana. Έχουμε αυτή την έκθεση τη πρωτοβουλία, αλλά σήμερα το πρωί είπαμε εγώ και οι σκιώδει ηγητέ ότι αντί να έχουμε την ε, διαδικασία αυτή, να χρησιμοποιήσουμε το έγγραφο εκείνο το οποίο εγώ ετοίμασα για την ε, ε, Οικονομική Επιτροπή και είπαμε ότι εκεί να προσθέσουμε τα, τα της εφαρμοστές νομοθεσίες και τα, τα, τα των τροπολογιών. Οπότε ε, να δώσουμε και άλλη μια διάσταση στην Επιτροπή μας. Έχουμε δύο ενημερωτικά πακέτα, έχουμε εκεί όλη την τεκμηρίωση που αφορά τις ε, χώρες του μνημονίου. Οπότε γι' αυτό και είπαμε στις αρχές του 2014 να γίνουν δύο μελέτες εις βάθος ε, για κάθε μία από αυτές τις τέσσερις χώρες του μνημόνιου. Αυτή είναι η διαδικασία. Βεβαίως, εμείς ασχολούμεθα με την πτυχή, την κοινωνική, την πτυχή της απασχόλησης. Δεν θα μιλήσουμε για τα θεσμικά ούτε για τα οικονομικά. Γιατί θα έχουμε εκθέσεις της ΕΚΟΝ και της ΑΦΚΟ πάνω στα θέματα που σας είπα. E Επίσης, θα ασχοληθούμε με τις τέσσερις χώρες του Μνημονίου Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος και Ιρλανδία. Δεν θα θίξει αυτή η έκθεση τις άλλες τέσσερις χώρες του Μνημονίου. Ισπανία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Λετωνία. Γιατί το πρόγραμμα της ε, Ισπανίας αφορά κάποια οικονομική αρρωγή και άλλες χώρες τρεις δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Οπότε το ισοζύγιο πληρωμών τους απλώς υποστηρίχτηκε. Άρα εκεί είχαμε διαφορετικές παρεμβάσεις. Τώρα μιλούμε για ολοκληρωτικές παρεμβάσεις στην οικονομία της χώρας. Για αυτές τις χώρες θα ασχοληθούμε. Για να δούμε τώρα την ε, ουσία και το σχέδιο κειμένου, το οποίο έχει τρία μέρη. Πρώτα-πρώτα έχουμε τα πραγματικά περιστατικά. Τα είναι γνωστά, αφορούν τις νομικές υποχρεώσεις όπως απορρέουν από τις συνθήκες, τις συνθήκες της Ένωσης αλλά και της διεθνείς στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ένωση. Καλύψουμε τον κοινωνικό χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης συζητήθηκε και θα συζητηθεί και στο μέλλον όσον αφορά την εφαρμογή του. Επίσης έχουμε και τις ε, υποχρεώσεις προς το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Στο δεύτερο τμήμα έχω αναλύσει πάλι κάποια πραγματικά περιστατικά και μετά θα συζητηθούν οι συνέπειες όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής το 2020. Είναι οι στόχοι γνωστοί. Το κοινοβούλιο τους έχει ασπαστεί. Μιλούμε βεβαίω πάντα για τον κίνδυνο για την φτώχεια, για τον αποκλεισμό, την αποτυχία όσον αφορά τη συμμετοχή στο σχολείο και την απασχόληση για αυτούς τους στόχους ε, του 2020 και καταλήγω σε κάποιες συστάσεις. Κατόπιν έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Τα έχετε εδώ όλα αυτά εγγράφως. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αναλυθεί ότι οι υποχρεώσεις πρέπει να ε, τηρηθούν και να δούμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Και για να μην κατέβουμε στην κόλαση όπως λένε οι ποιητές, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται το τι γράφει το άρθρο 9, διότι όλες οι πολιτικές σχεδρές Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να οδηγούν σε υψηλή απασχόληση, κατά πολέμηση του γενικού αποκλεισμού και στην κατοχή ζωοτροπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι υποχρεωτικά. Άρα θέλω να δω το κατά πόσον η εντολή της Τρόικα έλαβε υπόψη αυτές τις υποχρεώσεις ή εάν μείνουν στο χρονοτούλαβο. Και έχουμε το άρθρο 151 της Συνήθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα όσα επιτάσσει ο κοινωνικός χάρτης. Εκεί έχουμε το άρθρο 2 και το άρθρο 3. Αυτά βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ε, με την Σύνήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Τρόικα ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εκεί έχουμε στο άρθρο 28 τις συλλογικέ συμβάσει, στο άρθρο 30 έχουμε τι γίνεται όταν κανεί ε, είναι άνεργος, ε, το, το σύστημα διανοητική πρόνοια, το, το άρθρο 35 ε, για τις κρατικέ κοινοφελεί υπηρεσίες. Άρα, τι λένε οι δινείς μα υποχρεώσει, τι λένε οι συνθήκες. Και επίσης να δούμε από την άλλη μεριά, να δούμε εάν όλα αυτά καλύπτονται από το μνημόνιο. Επίσης, να δούμε κατά πόσο η Τρόικα έλαβε υπόψη τους στόχους του στρατηγής του 2020, δηλαδή απασχόληση, φτώχεια, αποκλεισμό από το σχολείο και κοινωνικό διάλογο έχουμε συζητήσει στην εκθεσή μου, αλλά καταλήξαμε ότι δεν έλαβε υπόψη η Τρόικα όλα αυτά. Δεν προέβη σε προηγουμένη ανάλυση. Τι έγινε επομένω με αυτές τις υποχρεώσεις, τις υποχρεωτικές υποχρεώσεις του ΣΥΠΗΝ. Και γι' αυτό έχουμε αρνητικέ συνέπειες. Ούτε έγινε κανένας είδους διαβούλευση με όλα όσα θεωρεί υποχρεωτικά σαν διαβούλευση Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ΟΚΕ, Επιτροπή των Περιφερειών, Επιτροπή Απασχόλησης, Κοινωνική Επιτροπή, τίποτε. Απλώς το Eurogroup αυτοί οι οποίοι συνέταξαν την εντολή της Τρόικας προχώρησαν σαν να μην υπήρχε τίποτα άλλο παρά μόνο τα χρηματοοικονομικά. Σαν να υπήρχε μόνο η χρηματοοικονομική πραγματικότητα. Τι έγινε, δεν να γίνει αλλιώς, παρά είδαμε πόσο έχει χτυπηθεί η απασχόληση. όχι μόνο δεν δημιουργήσαμε θέσει απασχόληση όπως λέει το στρατηγική 2020, αλλά φτάσαμε σε αρνητικό ρεκόρ καταστροφής, ε, ματέωσης, εξαφάνισης της συνεργασίας, που φτάσαμε στο 15%. Σε πολλές χώρες και σε ορισμένων κομμάτια του, του πληθυσμού φτάσαμε σε διπλασιασμό της ανεργίας μιλούμε για 50% της ανηλίας των νέων σε χώρες όπως η Ισπανία και επίσης πάρα πολύ δραματική κατάσταση σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως οι μετανάστες και οι γυναίκες. Φτάσαμε μέχρι το 20% κάτω από το μέσο Εκατομμύρια είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αυτά τα τρία χρόνια χάσανε τη δουλειά τους. Η ε, φτώχεια επίσης, εντυπωσιακά τα στοιχεία, το φορέα Κάρετα μας έχει κάνει μια έκθεση. Φτάσαμε και εδώ σε αρνητικά ρεκόρ. Και επίσης για τους ανήλικους έχουμε προβλήματα. Φτάσαμε 27% ε, για ανηλίκους που, που είναι κάτω από το κατόφυλλο της φτώχειας. Και το Συμβουλίο της Ευρώπης καταδίκασε τα σχετικά προγράμματα λόγω των συνεπειών τους και πρόκειται για κατάφορη παραβίαση του άρθρου 12 του Χάρτη και του άρθρου 4 του παρατήματος. Άρα, τίποτα δεν είναι για, το, για τους στόχους του 2020 και επίσης τίποτα δεν είναι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους νέους. Πάντως, είπαμε ότι κάθονται περισσότερο στην εκπαίδευση, ε, την εκούσια ή την υποχρεωτική, οι νέοι, γιατί δεν βρίσκουν δουλειά μετά. Επίσης ο κοινωνικός διάλογος και αυτός χτυπήθηκε, γκρεμίστηκαν δομές κοινωνικού διαλόγου, γυρίσαμε δεκάδες χρόνια στο παρελθόν, διαπίστωση αυτό και του διεθνούς Οργανισμού ή Γραφείου και επίση καταπατήθηκαν οι συλλογικέ συμβάσει. και έχουμε τώρα και ένα άλλο κεφάλαιο. Όσον αφορά αυτέ τι συστάσεις μου πρώτα πρώτα λέω ότι θα πρέπει να φωτιστεί πλήρω το σύνολο τη κατάσταση, όχι μόνο τα οικονομικά, τα μακροοικονομικά, αλλά θα πρέπει επιτέλους κάτι να υπάρξει που δεν υπάρχει όσον αφορά τα θύματα των αρνητικών συνεπειών της κατάστασης. Ζητήθηκε επομένω να κάνει μια αξιολόγηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι συνέβη. Υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες για να γίνει κάτι τέτοιο. Να ληφθεί υπόψη το 2020 και επομένω θα προκύψει ότι πρόκειται για μια τραγωδία. Δεν είναι η κατάσταση αυτή συγκυριακή. Είναι διαρθρωτική. Και η έχει πληγεί. Αυτά όλα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα αξιολογήσει και να υπάρξουν κάποια προγράμματα για οικονομική αρρωγή γιατί θα πρέπει να βοηθηθούν αυτές οι χώρες που χτυπήθηκαν από αυτή τη χώρα της ε, άκρατης βάρβαρης λιτότητας. Κάτι να κάνουμε για την ε, τρομερή αυτή φτώχεια που επικράτησε και καταστροφή του κοινωνικού ιστού και να μην επαναληφθούν οι τρόικες στο μέλλον. Δεν χρειαζόμαστε του Δουνουτου. Δεν χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Τράπεζα που να ενεργεί τελείως εκτός των ε, προβλεπομένων αρμοδιοτήτων της. Να δοθεί και από το Κοινοβούλιο και από όλους τους εμπλεγμένους μία απάντηση. Και έτσι, με αυτή την ευρωπαϊκή απάντηση, να ενεργήσουμε με αυτό, σύμφωνα με τις συνθήκες με αυτά τα 50 χρόνια της ευρωπαϊκής οικοδόμησης γιατί είναι σημαντικό να σώσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά πιο σημαντικό να σώσουμε τους νέους και τους ανήλικους που είναι το μέλλον της Ευρώπης. Με λίγα λόγια αυτή είναι η έκθεσή μου. Βεβαίως και θα πρέπει να αρθούν κάποια κοινά που υπάρχουν γιατί υπήρχε πίεση χρόνου, λίγος χώρος που έπρεπε να ενεργήσω όσον αφορά αυτές τέσσερις σύλλητες που έπρεπε να α, συντάξω και άρα θα πρέπει εμείς να συμπληρώσουμε το τοπίο όπως θα το διαμορφώσει η έκθεση της ΑΦΚΟ και της ΕΚΟΝ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική εκθέση για την Επιτροπή μας. Κάλλιο αργά παραποτέ, όπως λέμε, ε, γιατί είναι ζητήματα τα οποία καίνε το Κοινοβούλιο αυτά. Ευχαριστώ. Αρχίζει η συζήτηση τώρα. Καλό θα ήταν να ακούσουμε πρώτα πρώτα τους Κιώδης. Ρετζίνα Μπάστος, Μαρίαν Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλεχάνδρο Σέρκας για ε, την πλαισίωση της δουλειάς που έκανε για την έκθεση για τη δράση της Τρόικα στις ε, χώρες προγράμματος. Είναι πολύ καλά διαρθρωμένη η προσέγγιση που ακολουθεί Εξετάζει σφαιρικά λοιπόν τη δράση της Τρόικας σε αυτές τις χώρες και τις επιπτώσεις ε, αυτής της δράσης για τους επιμέρους στόχους ε, της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Δεν έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια αντίφαση σε σχέση με την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής μας ε, ως προς τις εργασίες της Επιτροπής ΕΚΟΝ και που έχει αναλάβει η Μαρίσα και έχει εντελώς διαφορετική δομή. Ε, πάντως ε, το πεδίο εφαρμογής ε, είναι πεδίο αρμοδιότητάς μας, απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, ε, ζητήματα που σχετίζονται με την φτώχεια, την εγκατάλειψη του σχολείου από τα παιδιά και ούτω καθεξής Αυτά συναποτελούν το πεδίο εφαρμογή της έκθεσης ε, του Αλεχάνδρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις τέσσερις χώρε προγράμματο ε, ε, απουσιάζει οποιαδήποτε δράση της Τρόικας σε, αυτό, σε, σε αυτούς τους τομείς που προανέφερα και περιορίζεται μόνο σε οικονομικά ζητήματα. Δηλαδή, η κατάσταση που βιώνουν αυτές οι χώρες και οι κυβερνήσεις ε, που ζήτησαν την παρέμβαση της Τρόικα ε, πρέπει να επομιστούν κάποιες ευθύνες. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ε, Ε, είναι μεγάλη σημασία των προγραμμάτων και των δανείων που εδόθησαν και των μέτρων που επιβλήθησαν ε, ούτως ώστε να είναι βιώσιμη η βοήθεια και ε, να συγκρίνουμε αυτή την κατάσταση που βίωσαν οι χώρες προγράμματος, οι χώρες μνημονίου, με την κατάσταση που θα υπήρχε αν δεν είχε υπάρξει παρέμβαση της Τρόικας σε αυτές τις χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε εάν ε, θα μπορούσε κάποια άλλη οντότητα, νομική οντότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαφορετική από την Τρόικα να ε, είχε παρέμβει αν δεν είχε ζητηθεί βοήθεια υπό αυτή την μορφή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δεν είχε εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο από, το, ε, από την Αγία Τριάδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εάν δεν είχε ζητηθεί αυτή η βοήθεια από τις χώρες ε, μνημονίου, ποιο θα ήταν το εναλλακτικό σενάριο. Θα πρέπει επίσης να δούμε σε ποιο βαθμό έχουν εφαρμοστεί αυτά τα, τα μέτρα και αν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Δεν πρέπει να θεωρείται τετελεσμένο γεγονός, δεν πρέπει ε, να θεωρείται ευκταία επανάληψη παρέμβασης, τέτοιου είδους παρέμβασης από πλευράς της Τρόικα σε άλλες χώρες που ενδεχομένως θα ζητήσουν βοήθεια με τρόπο ώστε να μπορέσουν ε, να συνεχίσουν ε, να έχουν χρηματοδότηση της διακυβέρνησης που έχουν αποφασίσει ε, και ε, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που έχουν επιλέξει. Αυτό είναι το θέμα μας. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ λύσεις ε, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναστροφή της κατάστασης σε σχέση με αυτή που έχει δημιουργηθεί στις χώρες μνημονίου. στην Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, μετά τις επισκέψεις που έγιναν σε αυτές τις χώρες, α, και να σας πω, ότι στις αρχές του 2014 έχει προβλεφθεί επίσκεψη στην Πορτογαλία. Έχουμε επίσης την ακρόαση των εμπειρογνωμόνων ε, στην ΕΚΟΝ, όπως και σε εμά εξάλλου ε, έχει προβλεφθεί να γίνει αυτό, πάλι στις αρχές του 2014 διότι το ζήτησαν πολλές πολιτικές ομάδες και θα έπρεπε ενδεχομένως να σκεφτούμε το ενδεχόμενο συνδυασμού των δραστηριοτήτων της ΕΚΟΝ με τις δικές μας. Ε, οι επισκέψεις στις χώρες μνημονίου θα έπρεπε να ενσωματώνουν στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τα προγράμματα της δική μας Επιτροπής, να μην ακολουθείτε μόνο το πρόγραμμα της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Πέρα από τις επιπτώσεις λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη πλαισίωση, ξαναλέω, για να κατανοήσουμε ποιε είναι οι ανάγκες αυτών των χωρών διότι σε αυτές τις ανάγκες βασίστηκε η αρχική ε, υποβολή ετοίματος για χορήγηση βοήθειας από την Τρόικα. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, ε, Μαριάν Χάρκιν και Ίνες ε, Τσούμπερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί ακόμα έχω πάρα πολύ δουλειά να κάνω για αυτή την έκθεση. Παρά το γεγονός ότι προέρχομαι από μια χώρα όπου είχαμε την παρουσία της Τρόικα ε, και μάλιστα την Κυριακή που μας πέρασε είχαμε μεγάλο ενθουσιασμό, γιορτάσαμε ε, το ότι έφυγαν από τη χώρα μας. Ε, βέβαια δεν μπορούμε να πούμε περασμένα, ξεχασμένα, κάθε άλλο. Θα ήθελα παρόλα αυτά να κάνω κάποια σχόλια. Εκτιμώ το γεγονός ότι η συγγήτρια άρχισε να κοιτάει τις ίδιες τις ε, συνθήκες και τα διάφορα άρθρα στις ε, συνθήκες και το πώς ακριβώς ε, υποτίθεται ότι αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Κυρίως το άρθρο υπαριθμών 9 και όπως σας είπα προηγουμένως και θα το ξαναπώ, ίσως να είμαι εδώ η μόνη βουλευτής η οποία είχε την ευκαιρία από κοινού με τους ε, συναδέλφους μου να πείσει τους Ιρλανδούς ε, πολίτες να υπερψηφίσουν τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Και αυτό κυρίως λόγω του άρθρου υπαριθμών 9. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον, για μένα τουλάχιστον, να διαπιστώσω κατά πόσον είχα δίκιο. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, άκουσα τι είπαν οι συνάδελφοι σχετικά με το ότι θα πρέπει να παραμείνουμε μέσα στις αρμοδιότητές μας. Κατανόητο αυτό, όμως όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020 πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτά εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας. Και θα ήθελα και πάλι ε, να κάνουμε μία σύγκριση. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Μπορούμε να μετρήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί ε, σε σχέση με το ποιοι ήταν οι στόχοι μας και επίσης μπορούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε άλλα κράτη-μέλη. Όπως ε, λοιπόν είπε και ο εισηγητής, ε, η μόνη περίπτωση όπου δεν υπάρχει αρνητική εξέλιξη είναι στους αποφύτους σχολείου, στην παιδεία. Οι άνθρωποι πριν από την πατρίδα μου έμειναν περισσότερο στα σχολεία γιατί δεν έβρισκαν δουλειά. Άκουσα και τι είπε η κυρία Μπάστας, ότι θα πρέπει να δούμε πού ακριβώς ξεκινήσαμε. Τα πράγματα είναι διαφορετικά βέβαια στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν θέλω πάλι να υπογραμμίσω την Ιρλανδική περίπτωση, αλλά ε, αν δούμε το ποσοστό του ΑΕΠ ε, το 7 ήταν 30% και κάθε χώρα ξεκίνησε από διαφορετικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια θα ήταν τα αποτελέσματα αν τελικά δεν είχε παρέμβει η Τρόικα. Δεν είμαι σίγουρη ότι πρέπει να το εξετάσουμε αυτό, αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν μπορούμε και να το αγνοήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν Καλό αυτό που υπάρχει αυτή η παρέμβαση. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Να σας πω, συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε ο εισηγητής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ε, ο δικός μας ο Επίτροπος ε, είναι λίγο κατηγορηματικός ε, στα σχόλια που κάνει και όταν μιλάμε για τις δραστηριότητες της Τρόικα, ένα από τα πράγματα που προσπαθούν να εστιάσουν την προσοχή τους είναι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας. Ο Επίτροπος ο ίδιος είπε ότι εστιάζουμε περισσότερο εκεί την προσοχή μας και όχι στην ε, πολιτική απασχόληση. Συμφωνώ. Εάν λοιπόν από όλα αυτά συνάγουμε κάτι, τότε είναι το να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε τώρα και να πούμε εντάξει, μέχρι τώρα αυτό είναι το αποτέλεσμα, θέλουμε να ε, συνεχιστεί η ίδια κατάσταση. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό το να κάνει κανείς μια έκθεση και μετά όμως πρέπει κανείς να διορτηθεί κατά πόσον αυτά επηρεάζουν κάτι ή απλά αν μιλάμε και μόνο στον εαυτό μας. Και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή για τη μέχρι τώρα δουλειά του. Ευχαριστώ Ίνες ε, Τσούπερ και Έντιτ ε, Στρέλα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή βάση για τις μελλοντικέ μας εργασίες αυτή που μας προσφέρει. Ε, ως επιτοπλίστων ε, συμφωνούμε για τη διάγνωση που κάνει είναι προφανές ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε, να βελτιώσουμε, να εμβαθύνουμε αυτή τη βάση για τις μελλοντικές μας εργασίες. Πέρα από την ιδιότητά μου ε, της σκιώδης για την QNGL, είμαι και Πορτογαλίδα και αυτό επηρεάζει τη συμβολή ε, που θα προσφέρω, τη συμβολή μου, διότι και εγώ βιώνω αυτή την πραγματικότητα καθημερινά. και αυτοί που, τους οποίους εκπροσωπώ επίσης. Ε, ζει η Πορτογαλία τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση στην ε, ιστορία της. 1,5 περίπου εκατομμύριο ανέργους έχει ε, και ένα μεγάλο ποσοστό ζει στο όριο της στόχιας, όπως αναφέρεται στην έκθεση. Έχουμε γυρίσει την δεκαετία του 50 ως προς την επενδυτική θέση της, θέση, της χώρας μας. Θα προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε τα θέματα της απασχόλησης από τα οικονομικά ζητήματα, αλλά θα καταλάβουμε πολύ σύντομα αν το αποπειραθούμε αυτό ότι είναι αλληλένδετα τα ζητήματα και δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Το ίδιο ισχύει και για τα κοινωνικά ζητήματα. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι η αυξανόμενη εκμετάλλευση των εργαζομένων ε, και η εκαθάριση των, δικαιωμάτων, των εργατικών δικαιωμάτων. Για το 2014 ο κρατικός προϋπολογισμός θα περικοπεί κατά 4,4 εκατομμύρια. Αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Τρόικα και θα σημάνει περαιτέρω περικοπές των μισθών και των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, των κρατικών ε, επιδομάτων, ε, των δημοσίων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, στον τομέα του πολιτισμού, ε, περικοπή των επιδομάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έτσι επηρεάζονται οι συνέργειες δημοσίου ιδιωτικού τομέα ε, και ε, τελικά συνειδητοποιούμε ότι προωθούνται ε, ιδιωτικά μόνο συμφέροντα μέσα από αυτά τα προγράμματα. Επίσης υποβάζονται τα δικαιώματα συλλογικής διαπραγματεύσης και διευκολύνονται οι μαζικές απολύσεις διευκολύνονται οι μαζικές απολύσεις ε, και με αυτόν τον τρόπο υποβιβάζεται η αρχική διαπραγματευτική θέση των εργαζομένων για την διαπραγμάτευση των βασικών τους μισθών. Επίσης, ε, αν συνδέσουμε αυτό το ζήτημα με το θέμα της ε, μετανάστευσης, ε, συνειδητοποιούμε ότι επηρεάζεται η αγορά εργασίας, διότι το 2013 130.000 εργαζόμενοι μετανάστευσαν, έφυγαν από τη χώρα. Η Πορτογαλία στη ζώνη ευρώ ήταν στην τρίτη θέση ως προς την αγοραστική δύναμη και την κατανάλωση ε, πριν ε, την κρίση. Βλέπετε λοιπόν ότι τώρα με τη γενικευμένη πτώχευση της ε, χώρας, τον αρνητικό αντίκτυπο των μέτρων στους εργαζόμενους, διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε αντιμετωπίσουμε και την αποκρατικοποίηση του ταχυδρομείου στην Πορτογαλία και ε, από ό,τι προβλέπεται στο μνημόνιο ο αερομεταφορέας Πορτογαλίας, η ΤΑΠ, ε, θα ακολουθήσει. Αυτό θα επηρεάσει, ε, θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση ως προς τις απολύσεις και την αγοραστική δύναμη των Πορτογάλων. Πάντως ε, το μεγαλύτερο ζήτημα είναι πολιτικού χαρακτήρα. Ποια, πώς νομιμοποιείται η Τρόικα για να επιβάλλει τέτοιες ε, επιλογές ε, που αντίκειται στις κυρίαρχες αποφάσεις των κρατών και αντίκειται κυρίως στη δημοκρατική βούληση των πολιτών των χωρών αυτών. Βεβαίως αυτό το ζήτημα ίσως να απασχολήσει περισσότερο την ΑΦΚΟ και όχι τη δική μας Επιτροπή. Θέλω να σας ε, ε, να αναφέρω ότι συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι είναι η λογική ε, της Τρόικας συνάδει με τη λογική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δρά στην ε, Λατινική Αμερική και είδαμε τα καταστροφικά αποτελέσματα της δράσης. Βλέπουμε λοιπόν, κάνουμε τη σύγκριση και οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η λογική της Τρόικα ακολουθεί την ίδια ρότα και θα πρέπει να ε, επαναδιαπραγματευτούμε τα χρέη με τους δανειστές μας, ε, διότι σήμερα πλέον είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να ε, προσαρμόζεται το ύψος του δανείου στη στα οικονομικά αποτελέσματα της ε, χώρας και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας αν υπάρχει. Εγώ δεν ξέρω τίποτα από οικονομικά ζητήματα, μου φαίνεται προφανές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο. Πρόεδρος Εντίτε Στρέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή μας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνει και συμμερίζομαι τις ανησυχίες του. Θεωρώ ότι η κοινωνική διάσταση είναι ε, κέρια σημασία σε μια έκθεση τέτοιας φύσης. Θα ήταν ανήκουστο να γίνει αξιολόγηση των επιπτώσεων των μνημονίων που εφαρμόζει, που επιβάλλει θα έλεγα μάλλον η Τρόικα χωρίς ε, να προσδώσουμε ε, την δέουσα σημασία στην κοινωνική διάσταση και στο κοινωνικό κράτος ε, όπου είναι πλέον προφανείς οι αρνητικές επιπτώσεις των νημονίων. Ήδη είπε ο εισηγητής αλλά και άλλοι συνάδελφοι μιλώντας για το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού, της αυξησιστής της της ε, όξυνσης των ε, κοινωνικών ανισοτήτων, της αύξησης ανεργίας των νέων. Ε, α, και να πω εγώ παρενθετικά πως σημειώνεται μια επίθεση κατά της μεσαίας τάξης. Θυσιάζεται η μεσαία τάξη στο βωμό των πολιτικών των κυβερνήσεων και των προγραμμάτων που ε, επιβάλλει η Τρόικα για όσους παρατηρούν, παρατηρούν την κατάσταση απ' έξω ε, ίσως δεν είναι ε, προφανές αυτό δεν είναι προφανές να γίνει η διάκριση ανάμεσα σε αυτά που επιτάσσει η Τρόικα και αυτά που επιθυμούν ε, οι κυβερνήσεις διότι ορίζονται κάποιοι στόχοι αλλά σίγουρα δεν υπάρχουν μονόδρομοι για να επιτευχθούν ε, οι προκαθορισμένοι στόχοι. Λοιπόν, ε, υπάρχει μη ένας υπερθεματισμός ε, ως προς την λιτότητα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ταυτόχρονα η δημιουργία, η απαραίτητη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η απαιτούμενη οικονομική μεγέθυνση. Δεν αντιλαμβανόμαστε πώς ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ευρωπαϊκών ηθινόντων ή σε εθνικό επίπεδο δεν λαμβάνονται υπόψη ε, οι γνωμοδοτήσεις ε, ε, που προέρχονται από νομπελίστες οικονομολόγους οι οποίοι μας διαβεβαιώνουν ότι είναι υπερβάλλουσα η λιτότητα και ότι θα έχει καταστρεφτικές συνόπειες για τις επερχόμενες δεκαετίες η λιτότητα δεν έλυσε κανένα από τα προβλήματα και το αντίθετο δημιούργησε νέα προβλήματα, διευρύνοντας και το χάσμα ε, ανάμεσα στους πλουσίους και τους φτωχούς, ε, τους έχοντες και τους μη έχοντες ε, στη χώρα μου, κάτι που μας καταπλήσει. Κάποιους από εμά οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι και ε, προέκυψαν ε, φύτρωσαν σαν μανιτάρια 25 νέοι εκατομμυριούχοι στην Πορτογαλία. σε σχέση με την ε, έναρξη του μνημονίου. Αυτό θα πρέπει να αναφερθεί επίσης δράση της Τρόικα δεν πρέπει να παραβιάσει συνταγματικές αρχές. Ε, δηλαδή, η χρηματοδότηση είναι συνάρτηση εφαρμογής προκαθορισμένων πολιτικών. Ε, το τεστ είναι επιβολή ενός συγκεκριμένου κοινωνικού μοντέλου που ε, οδηγεί σε μετουσίωση του κοινωνικού κράτους, σε εκφυλισμό του, ε, σε ένα κράτος φτωχών. Είναι υπαρξιακό πλέον το ζήτημα. Ε, αλλάζει, εκφυλίζεται, ξαναλέω, το κοινωνικό κράτος και η πολιτικές έχουν καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο στο κοινωνικό κράτος αλλά και στον τομέα της υγείας. Αυτά είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του εκφυλισμού η Τρόικα και οι οντότητες που υπάρχουν πίσω από την Τρόικα και χρηματοδοτούν γνωρίζουν την κατάσταση και ε, κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά από τα δάνεια. Παράδειγμα τους χάρη, η Πορτογαλία ε, στην αποπληρωμή του χρέους δάπανα ε, ποσό ε, αντίστοιχο με τις περικοπές των κοινωνικών δαπανών. Ο Ζώζ Αταλή ε, και άλλοι δεν αναφέρθηκαν στην Πορτογαλία βέβαια, αλλά ε, γενικότερες χώρες μνημονίου είπαν ότι ε, δύο είναι τα τεινά για τους νέους. Ή θα εγκαταλείψουν τις χώρες τους ή θα ξεκινήσουν μία επανάσταση. Κατά πάσα ε, πιθανότητα θα πρέπει να τους ζητήσουμε να δράσουν και άρα να επαναστατήσουν μέχρι ότου κάποιος επιτέλους να δώσει ε, σημασία στο μέλλον των νέων, γιατί ε, αν δεν έχουν μέλλον οι νέοι και συνειδητοποιήσουν ότι τα όνειρά τους μετατρέπονται σε εφιάλτες, ε, καταλαβαίνετε ότι θα οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις που πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Karine Mandeli και ε, Εύελιν Ρέγνερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να σα ευχαριστήσουμε πρώτα πρώτα εσάς, διότι η έκθεση αυτή τη πρωτοβουλία είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία σε μία περίοδο που είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κανεί τον αποτυπωμπαίο τράγο στην Ευρώπη. Οπότε και έχουμε την εντύπωση ότι όλο ένα και πιο σπάνια ακούμε καλά μαντάτα. Όμως είναι καλό μαντάτο αυτή η έκθεση. Μπράβο κύριε Θέρκα, ευχαριστούμε. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε να φανεί ότι αυτές οι χώρες είναι αποκοτευμένες, αλλά το αντίθετο, ότι ξεπηδάει μια καινούργια δυναμική, γιατί ναι, υπήρξαν ε, λάθη όσον αφορά την επιβολή της λιτότητος. Πολλά θα πρέπει να γίνουν, αλλά θα πρέπει πρώτα-πρώτα να εγκαταλείψουμε αυτή τη λογική. Κάθε μιλούμε για τρόικα, έχουμε κατά νου το ότι θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να σφίξουν περισσότερο το ζωνάρι τα επόμενα χρόνια. Και ότι οι προϋπολογισμοί πρόκειται να περικοπούν ακόμη περισσότερο κυρίως όσον αφορά τις κοινωνικές τους δαπάνες. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο, χάσμα μεταξύ αυτών που θα ωφεληθούν από αυτή την επανεκκίνηση και των λοιπόν. Εκείνων δηλαδή που ακόμα δεν έχουν μπει στην ρότα της επανεκκίνησης. Και εγώ στο κείμενό μου στάθηκα σε διαφορά σημεία. ασχολήθηκα με τα κοινωνικά θέματα και όχι με τις φούσκες της αγοράς των ακινήτων. Όταν η Τρόικα ζητάει να γίνουν δαπάνες, μιλάμε για στεγαστικά δάνεια. Χιλιάδες. Για να πληρώσουν τα δάνεια αυτά, μένουν στο δρόμο. Άστεγες πολλές οικογένειες. Επίσης, η επασχόληση ένα σημείο εις το οποίο θα πρέπει να υπόψη τις εκθέσεις μας το τι, θα, τι έγινε και τι θα γίνει τι θα γίνει σε σχέση με το περιβάλλον και την ενεργειακή πολιτική θα πρέπει εδώ να διατυπώσουμε κάποιες έντονες συστάσεις γιατί μιλούμε για κάποιους κλάδους που αντιστέκονται στην κρίση. Μιλάμε για την οικονομία της ελληνικής, οπότε θα πρέπει να επαναεκβιομηχανίσουμε ούτως υπήν την Ευρώπη. Να το πούμε αυτό. Επίσης, ένα το ερώτημα το τι θα γίνει όσον αφορά τις κοινωνικέ επενδύσεις. Και ρωτώ με το κείμενό μου, εάν ζητούσαμε από την Επιτροπή να συντάξει μια έκθεση. Αν γινόντουσαν όλες οι σχετικές κοινωνικές επενδύσεις μέσα στην κρίση. Δεν θα πήγαινε καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, μην ανησυχείτε από μένα, θα ακούσετε μία και μόνο πρόταση. Ο κύριος Κάρας είπε σήμερα ότι η Τρόικα είναι έσχατη λύση έσχατη λύση για πολιτικές ε, έκτακτες καταστάσεις. Ακόμα και μια τέτοια λύση ποτέ δεν δικαιολογεί την παραβίαση κοινωνικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο Αλεχάνδρο το είπε με πολύ εντυπωσιακό τρόπο και γι' αυτό το λόγο τον ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή του. Ευχαριστώ. Θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Οπότε, ο συγκεκριτής μας να ολοκληρώσει. Λυπάμαι που δεν έχει να πει κάτι η Επιτροπή μας, αλλά μετά από τρία χρόνια, το ότι δεν είπε κάτι η Επιτροπή Ευρωπαϊκή είναι ακόμα χειρότερο. Δεν θα πρέπει όλα αυτά να τα έχετε συζητήσει, να τα έχετε πει για το Δούνε για την Κεντρική Τράπεζα, για το Eurogroup που έχει γίνει κάτι σαν διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Διαβάστε το μνημόνιο. Κοιτάξτε τι έγινε με τους δανειστές. Τους έλειψε η ανθρωπιά. Συνάδελφοι, όπως και εσείς, έχω και εγώ να διαπιστώσω ε, τα ίδια, σας συγχαίρω, σας ευχαριστώ και πρόκειται κατά το έργο μου να λάβω υπόψη όλα όσα είπατε. Όλα όσα είπατε είναι πάρα πολύ εύστοχα. Θα πρέπει κάποια πράγματα να τα ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Γιατί είναι αλήθεια ότι όλοι έχουμε την αίσθηση ότι το ότι έχουμε συναρμόδιες τρεις επιτροπές αυτό δεν μας αφήνει να δούμε το θέμα σφαιρικά. Εμείς τώρα προσπαθούμε να σώσουμε από κοινωνική πτυχή σε αυτό το θέμα. Όπως το είπε η Εστρέλα, να αναλύσουμε τις ε, κοινωνικές συνέπειες, αλλά έχουμε τρεις άνθρωπες επιτροπές. Όπως είπε η Μπάστος, το χρέος, το έλλειμμα, προβληματική για το τι κάνουμε την κρίση. Έχουμε την ΑΦΚΟ, έχουμε την ε, οικονομική που ασχολούνται με τα δικά τους θέματα. και ε, καλά, δεν μπορεί κανείς να μείνει σιωπηλός ενώπιον αυτών. Δεν θα ήταν τόσο έξυπνο αν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα κοινωνικά. Άρα, θα πρέπει να συζητήσουμε με δημιουργικό τρόπο, παραγωγικό. Και μπορεί να βρεθεί συνένεση για τα κοινωνικά. Άρα, για να αποφύγουμε τα ίδια στο μέλλον, να αντλήσουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Προσοχή με των τροπολογιών για να περιοριστούμε στις κοινωνικές συνέπειες, τις συνέπειες της απασχόλησης σε αυτές τις τέσσερις χώρες γιατί μιλούμε τώρα για τα προγράμματα, για τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τις πολιτικές των κυβερνήσεων των πρώτων αυτών, γιατί αυτές οι χώρες υποχρεώθηκαν να κάνουν αυτά που κάνουν. Ε, διαβάστε λοιπόν το μνημόνιο. Το Central Europeo, que tienen otros mandatos en los tratados, dicen cómo tiene que ser la ley de arrendamientos rústicos o cómo tienen que ser cuestiones en las que ellos, tan celosos de su independencia. Γιατί ε, κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να αφήσουμε περιθώρια σε αυτές τις χώρες να πετύχουν τους στόχους τους αλλά με ανεξαρτησία. Προσπάθησαν να προσαρμοστούν σε αυτές τις πολιτικές που επιβλήθηκαν στη χώρα τους. Μιλάμε για κάποια, ε, κάποιους κανόνες που παραβαίνουν το Σύνταγμα μιας χώρας όπως την Πορτογαλία και γι' αυτό και το Συνταγματικό Δικαστήριο εκήρυξε τα μέτρα αντισυνταγματικά. Ρετζίνα, δεν θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε το ότι η οικονομική κατάσταση επέβαλε τέτοια αντιμετώπιση. Εγώ νομίζω ότι χρειαζόντουσαν κάποια προγράμματα, αλλά το θέμα είναι τι είδους προγράμματα θα ήταν. Δηλαδή, ναι, να χορηγηθεί βοήθεια, αλλά υπό ποιες προϋποθέσεις. δεν ήταν δυνατόν να δοθεί τέτοιο χτύπημα στα προγράμματα, στις πολιτικές του κράτους προνοίας. Το αντίθετο, αυτά θα έπρεπε να διασωθούν. Τα ανάειλησε αυτά το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και παρέπεμψε στην, στο θεμελιώδη χάρτη δικαιωμάτων που σε θεμελιώδη σημεία του κατεπατήθηκε. δεν θα έπρεπε στο βωμό της ε, επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων να καταπατηθούν τόσο και τόσα. Τίποτα δεν έκανε η Τρόικα για να προβλέψει τις συνέπειες των ενεργειών. Γιατί σε τόσες και τόσες σελίδες μνημονίου ή μνημονίων δεν υπάρχει ούτε κεραία για αυτούς όλους τους φτωχούς. Ο κύριος Ολιρέν υπέγραψε αυτά τα μνημόνια και θα μείνει στην ιστορία για αυτό το οποίο έκανε. Κύριε Χάρκιν, επίση. συμφωνώ μαζί σας. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών επίσης με εκπλήσει και αυτό. Υπάρχει, είδατε, συμμετρία, παραλληλισμός των ε, των, ε, των, των μέτρων που επιβλήθηκαν. Όμως το καθένα είχε άλλο είχε άλλα προβλήματα το καθένα κράτος. Όμως πρέτα ποτέ στους ψηλού, στους κοντούς, στους, χοντρού, χοντρούς, στους αδύναμους, όλοι, όλοι στο, στο, στο, ίδιο μοντέλο χωρέσαμε. Για συντάξεις, για παραγωγή, όλα. Τα λέει αυτά. Α, στι συντάξει στην Ισπανία. Είχαμε 60 δις πλεόνασμα και όμως μας υπευλήθησαν τα ίδια μέτρα όπως σε χώρες που είχαν τρομερό έλλειμμα. Άρα, είχαν στο μυαλό τους τα οικονομικά προβλήματα και όχι τον κόσμο εις τον οποίο θα επιβάλλονται αυτά τα μέτρα. Εντάξει, συμφωνώ όπως λέει η κυρία Βάστος, το θέμα δεν είναι τώρα να, να κλαίμε ό,τι έγινε έγινε, να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον και επίσης να δούμε το πώς θα μάθουμε τα, μάθημα, τα λάθη και στο μέλλον θα κάνουμε τα ίδια εναλλακτική και στις συστάσεις αυτό λέω ευρωπαϊκό πρόγραμμα να γίνει και όχι όπως τώρα το οποίο είναι τελείως έξω να καταπολεμήσουμε τις ασυμμετρίες τα μακροοικονομικά προβλήματα των χωρών, να διορθωθούν τα κουσούρια του χρηματοοικονομικού ε, του χρηματοοικονομικού συστήματος να σταματήσουν οι, τα φυσικά πρόσωπα να πληρώνουν τις αμαρτίες του κρατικού προπολογισμού. Επομένως, το θέμα δεν είναι το να υπάρχουν δανειστέ και οι οφειλέτε. Είμαστε άνθρωποι, άνθρωποι και δεν είναι δυνατόν αυτοί με τα σκούρα κουστούμια να πηγαίνουν και να κλείνουν τα νοσοκομεία. Έχουμε όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία λόγω ελλημάτων και χρέους, όλα αυτά επιβλήθηκαν. Όμως έγιναν και άλλα πολλά ότι δηλαδή πέρα από τα οικονομικά προβλήματα και με, τη, με αυτή την πρόφαση εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους οι λεγόμενοι δανειστές για να καταστρέψουν κατακτήσεις δεκαετιών. Περιμένω επομένω τις ε, τροπολογίες σας, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί που σας είπα. Άρα έτσι να κάνουμε τη διάγνωση του τι έγινε και επίσης να δούμε πώς δεν θα ξαναγίνουν όλες αυτές οι, όλα αυτά τα φρικτά λάθη και στο μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Σίτα. Καταλαβαίνω την έκκληση που απευθύνεται όλοι να σεβαστούν ε, το φάσμα των αρμιδιοτήτων της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ε, Πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποια ζητήματα που σχετίζονται με την μεθοδολογία και όχι με την αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Ε, Φερρυπίν, ε, πολλά και καταδικάσαμε είτε τη δράση της Τρόικα είτε ε, εκφράσαμε τη θλίψη μας ε, που δεν συνδέεται στις εργασίες η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και την αντικαθιστά η Τρόικα. Αυτό, τέτοιου είδου ζητήματα νομίζω μπορούμε να τα εγείρουμε στι τροπολογίε. Πέραν αυτού, ε, ω προ την συγγήτρια της επιτροπή ΕΚΟΝ, ε, έχουμε κάθε συμφέρον να υπενθυμίσουμε ότι στην αρχή τη θητεία του το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο σε μια έκθεση για την οποία ήμουν εγώ αρμόδια, ε, ειδική έκθεση για την κρίση, αυτό ήταν ο τίτλο, είχε ορίσει ένα διαφορετικό σενάριο, χάρη στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εξέλθει από αυτήν την κρίση και την απόκληση των ε, οικονομιών με πολύ καλύτερο τρόπο αντί να βυθιστεί με στην ύφεση λόγω ε, των πολιτικών ε, λιτότητες που έπληξαν τις ασθενέστερες οικονομίες της Ένωσης. Λοιπόν, αυτό νομίζω πρέπει να φανεί επίσης μέσα στις τροπολογίες μας δεν ε, μιλήσαμε για ένα τεχνικό ζήτημα. Ε, συντάξατε το σχέδιο γνωμοδότησης ως ε, γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ΕΚΟΝ και δικαίως λόγω έλλειψης χρόνου δεν καταθέσατε ε, νέο σχέδιο, απλώς θα το μεταμορφώσετε σε έκθεση πρωτοβουλίας. Όμως ε, τίθεται ζήτημα ε, για την αιτιολογική σκέψη πλέον. Καταλαβαίνω ότι έχετε ένα σχέδιο υπομάλης, ας το πω έτσι, και εδώ παραπέμπω και στην κοινή ακρόαση με την Επιτροπή έκων για την Ελλάδα. Ε, κατόπιν εντολή τη διάσκεψης του Προέδρου, νομίζω πρέπει να το υπενθυμίσουμε, μόνο και μόνο για να θυμίσουμε ότι έπρεπε να, να συμμετάσχουμε και εμείς κανονικά, τέλος πάντων. Το λέω διότι καταλαβαίνω ότι αυτές οι αιτιολογικές σκέψεις θα τις υποβάλλετε ε, υπό τη μορφή τροπολογιών προς τη δική σας έκθεση. Ε, ε, μπορείτε να μας, παρότι τα έχετε μόνο στα αγγλικά προς το παρόν όπως και την υπόλοιπη έκθεση, να τα δώσετε λοιπόν ήδη στους συναδέλφους ούτω ώστε να έχουν χρόνο αν θέλουν να καταθέσουν τροπολογίες και να συμβάλλουν στην έκθεση πρωτοβουλίας πλέον. Έτσι. Για το κομμάτι αιτιολογικέ σκέψει. Εκτός αν υπάρχουν ενστάσει, δεν υπάρχουν. Πολύ ωραία το αποφασίζουμε. και ε, θα ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι με ε, email για να είναι ξεκάθαρη ε, η διαδικασία. Λοιπόν, για τις τροπολογίες θα έχουμε μια γενναιόδορη προθεσμία για τις τροπολογίες. Ε, θα έχετε χρόνο να δουλέψετε για τη διάρκεια των διακοπών σας. Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου ε, ε, ε στις 12 ε, στις 3 Φεβρουαρίου θα τις εξετάσουμε τις τροπολογίες, τις συμβαστικές θα τις εξετάσουμε στις 12 Φεβρουαρίου και θα ψηφίσουμε την επόμενη μέρα στην Επιτροπή Απασχόλησης, ε, δηλαδή στις 13 Φεβρουαρίου και στην Ολομέλεια θα φτάσει το Μάρτιο η έκθεση. Εκ παραλίλου φαντάζομαι με τις εργασίες που θα γίνουν στην Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, υπό την αιγίδα των δύο συνεισηγητών. Ε, ελπίζω να μπορέσουμε να ακούσουμε και ε, κάποιους ε, εμπειρογνώμονες για τα όσα διακυβεύονται στο μεταξύ. Από ό,τι κατάλαβα η ΕΚΟΝ θα οργανώσει και μια ειδική ακρόαση ούτως ώστε να εισακουστούν και οι κοινωνικοί εταίροι. Εάν αυτό ισχύει, είναι προφανές πως θα ζητήσουμε κι εμείς να ε, οργανωθεί από κοινού τουλάχιστον αυτή η ακρόαση εφόσον πρόκειται για κοινωνικούς εταίρους. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις... Α, συγγνώμη, παρακαλώ. Κύριε Σέρκας. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ενημερώσω τους τη Επιτροπής και όλους όσους μας ακούνε από το διαδίκτυο ότι το Κοινοβούλιο έχει στο LinkedIn ανοίξει μια ομάδα ζήτησης για αυτή την έκθεση στο οποίο είναι πρόσβαση, στο οποίο ε, έχει πρόσβαση όποιος θέλει να συμβάλλει. Alors, euh, comme euh, le la Commission de l'emploi et des affaires sociales est à la pointe de... Είμαστε στην αιχμή της κοινωνικής καινοτομία εδώ στην Επιτροπή Απασχόληση. Λοιπόν, θα είμαστε και στην αιχμή της ε, δημοκρατικής καινοτομίας. Ε, έχουμε δρομολογήσει πιλωτικό πρόγραμμα ε, του οποίου η υλοποίηση θα πάρει σάρκα και ωστά μέσα στην έκθεσή σας. Είναι μεγάλη προσθεμένη αξία για το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, θα είστε στο Κέσαρα της Επιτροπής ε, Απασχόλησης ως προς την ε, καινοτομία. Μέσα στην έκθεση υπάρχει και διαδικτυακός ε, σύνδεσμος, ώστε με την αναμετάδοση στο διαδίκτυο να συμβάλλουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν και με την συμβολή τους, και συμβολή τους ελπίζω να μετατραπεί σε ε, συγκεκριμένα στοιχεία που θα συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας. Λοιπόν, τώρα θα ασχοληθούμε με το μεγάλο πακέτο των απαλλαγών. Ε, για τις πέντε εκθέσεις ε, προτείνω κοινή συζήτηση να γίνει απαλλαγή για το Γενικό Προϋπολογισμό πρώτα απ' όλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την ασφάλεια, την υγεία, για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση Συνθήκων Διαβίωσης και εργασία, στην ανάπτυξη τη επαγγελματική κατάσταση εντεφό, ε, το γενικό πλαίσιο είναι προφανές, ε, σχετίζεται με την ολοκλήρωση των εργασιών του ελεγκτικού συνεδρίου ως ε, προς ε, το κλείσιμο των προϋπολογισμών του προηγούμενου έτους, του 2012. Είναι προφανές ότι το ελεγκτικό συνέδριο θεώρησε ότι έγιναν διάφορα σφάλματα ως προς ε, τον ε, οικονομικό έλεγχο ε, των ε, δαπανών και ότι ήταν εν μέρει αποτελεσματική η οικονομική έλεγχη που έγιναν. Για το 2012 συγκεκριμένα αυξήθηκαν συνολικά τα λάθη ε, που εντοπίστηκαν ως προς τις πληρωμές. Το ποσοστό από 3,9 αυξήθηκε σε 4,8% και για τις κοινωνικές υποθέσεις ειδικότερα είναι καλύτερα η κατάσταση. Παρ' αυτά αυξήθηκε το ποσοστό των σφαλμάτων διότι από το 2,2 ε, είμαστε πλέον στο 3,2 μια ποσοστία μονάδα αύξηση δηλαδή. Για το παιδί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Απασχόλησης. Μιλάμε ουσιαστικά για τα κονδύλια του ΕΚΤ. Διότι από εκεί προέρχονται το 97% των δαπανών ε, που σχετίζονται με την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις. Αυτά ισχύουν για το 12. Οι υπόλοιπε δαπάνες είναι δαπάνες ε, που ε, πολύ σε χρηματοδοτούνται από επιδοτήσεις και ενισχύσεις που έχουν χορηγήσει οι αρμόδιοι οργανισμοί. Η βασική κίνδυνη που εντοπίζει το ελεγκτικό συνέδριο σε σχέση με τις δαπάνες για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σχετίζονται με τον άειλο χαρακτήρα των δαπανών, ε, μιλώντας για επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως ε, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή δυνατότητες συγχρηματοδότηση ε, για την απασχόληση πολλών κοινωνικών εταίρων. Αυτά μας οδηγούν ε, σε μεγαλύτερες δυσκολίες, αλλά αιτιολογούνται από τη φύση των ε, δράσεων που έχουν αναλυθεί στο κοινωνικό τομέα. Αυτή η πολιτική εξετάστηκε και ελέγχθηκε ε, με τρόπο ε, εν μέρει αποτελεσματικό και σας είπα ότι για την περίοδο του 2012-2013 ε, το ποσοστό λάθους κυμαίνεται στο 3,2%. Ε, σας υπενθυμίζω τα πορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου τους ώστε να είναι πλήρως διαφανές το πλαίσιο στο οποίο θα συζητήσουμε τις απαλλαγές. αυτά Ε, αυτές τις αδυναμίες εντοπίζει το ελεγκτικό συνέδριο ε, μετά την ε, εξέταση των αιτήσεων. Εγώ δεν νομίζω ότι θα συμφωνούσαν ε, όσοι εφαρμόζουν τις δια, τα προγράμματα που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τέλο πάντων αυτά αποφάνθηκε το ελεγκτικό συνέδριο. Τα ή κανόνες επιλεξιμότητας σε εθνικό επίπεδο επίσης θα πρέπει να εξεταστούν ε, κατά τη γνώμη του ελεκτικού συνεδρίου για να ε, διαπιστωθεί αν ε, είναι δυνατή κάποια απλούστευση διότι η περιπλοκότητα των κανόνων οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού λαθών και ζητά ή δυνατόν απλούστευση των κανόνων. Ζητά επίσης να προαχθεί η χρήση απλουστευμένων κανόνων όπως μόλις σας είπα διότι αυτό ελαχιστοποιεί το ποσοστό λάθος. Ε, για τις νομοδοτήσεις για τις απαλλαγές, εκεί αναφερόμαστε διάφορες γνώστες ανησυχίες πιο συγκεκριμένα. η εποπτεία και ο έλεγχος ε, του βασικού εργαλείου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να ευθυγραμμίσετε πλήρως με τους στόχους πολιτικής Ευρώπη 2020 και φυσικότερα με το συνολικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, η γνωμοδότηση που υποβάλλεται προς έγκριση ζητά επίσης να εγκριθούν διάφορες προτάσεις ώστε να ε, μειωθεί έτσι περαιτέρω το ποσοστό λαθών ε, και χαιρετίζει τη δρομοέναρξη του προγράμματος Your First Job ε, που ε, συνιστά ρηξικέλευτη δράση και προτείνει και προσαρμογή του μηχανισμού ελέγχου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας για τους Απόρους ούτως ώστε να διαπιστώσουμε ε, ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζονται ε, οι ίδιες ε, προδιαγραφές ελέγχου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αφενός και αφετέρου για το Ταμείο Βοήθειας για τους Απόλους. Ως προς τους εξωτερικούς οργανισμούς τώρα, συνολικά για το 2012 αυτοί οι οργανισμοί συμμορφώθηκαν με, τις, με το προαπαιτούμενο ως προς τις διαδικασίες οι οποίες ήταν νομότυπες για το το ΣΕΝΤΕΦΟΠ στη Θεσσαλονίκη προτείνουμε ε, να επικροτήσουμε επιτέλους τον διορισμό ε, του Διευθυντή στο ε, Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτασης στο Τωρίνο. Εγκρίνουμε ε, τα μέτρα που ελήφθησαν για να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του ιστορικού, οι ιστορικοί λογαριασμοί μάλλον του εξωτερικού αυτού οργανισμού. Ε, εγκρίθηκαν νέε μέθοδοι για την πρόσληψη προσωπικού, τι οποίες επίσης επικροτούμε. όλα αυτά, προσοχή για το 2013, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει δυσκολία παρότι ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ανανεώθηκε η θητεία της Μανίλα Σερμπάνε, της Διευθύντριας, παρόλα αυτά η διαδικασία που εφαρμόστηκε ως προς τη διαθεσμική συμφωνία για το διορισμό διευθυντών εξωτερικών οργανισμών καθώς και σε σχέση με το ιστορικό καταστατικό του οργανισμού δεν ήταν ομότυπη η διαδικασία διότι δεν μας ζητήθηκε διαβούλευση και παρότι χαιρόμαστε για τον επαναδιορισμό της εφόσον μιλάμε το 2013 θα έπρεπε να μας έχουν διαβουλευτεί ε, και το αναφέρουμε, το τονίζουμε αυτό. Και παρόλα αυτά ζητάμε να χορηγηθεί ε, η απαλλαγή. Για το ETF... Ζητάμε να ε, ε, ε, εγκρίνουμε την συμφωνία για τη νέα έδρα του οργανισμού. Για τον επόμενο οργανισμό με έδρα το Δουβλίνο βλέπουμε μεγάλες μεταφορές κονδυλίων διότι υπήρχαν ε, μη προγραμματισμένες εργασίες. Αυτό πάντοτε αποτελεί κόλλημα για την ορθή εφαρμογή ενός προγράμματος εργασίας. Για τον τέταρτο οργανισμό, ε, όσα ε, ασφάλεια στον τομέα της υγείας, στο Μπιλμπάο, βρέθη και εκεί η έδρα. Πρέπει να κάνουμε όμως μια παρατήρηση διότι επιδέχεται βελτίωση ο τρόπος με τον οποίο διεκπεραιώνονται οι διαγωνισμοί. Η προτάση υποβολής πυροπροσφόρων. Για ε, την οικονομική διαχείριση σας προτείνω να αναφέρουμε ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ως ε, αρμόδια επιτροπή να γίνεται συζήτηση ε, για τους αιτήσεις λογαριασμούς. Λοιπόν, σας προτείνω να γίνει κοινή συζήτηση για τις πέντε αυτές απαλλαγές. Παρακαλώ ποιος θέλει το λόγο. Non, Marianne η κυρία Χάρκιν. Κυρία Πρόεδρε, τα είπατε όλα, δεν αφήσατε τίποτα. Τι να πούμε κι εμείς, είπατε τα περισσότερα από αυτά που μπορεί κανείς να πει. Και το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι σε σχέση με την απαλλαγή πιστεύω ότι η πρότασή σας στην παράγραφο 3 εκεί όπου του 2012, εκεί αναφέρομαι. Όχι, δεν αναφέρομαι στην, ε, στον οργανισμό, αναφέρομαι στην Επιτροπή. Μιλάτε για τα διάφορα εργαλεία, για το κοινωνικό ταμείο, τις μικροχρηματοδοτήσεις ε, θα πρέπει να διευκρινίσουμε λιγάκι σε σχέση με τους στόχους του 2020 και αυτό είναι χρήσιμο, πρέπει να το κάνουμε. Πριν από λίγο μιλήσαμε για τους στόχους, άρα δηλαδή πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε. Επίσης, άκουσα όλα αυτά που είπατε σχετικά με τους ε, βασικούς κινδύνους ε, με βάση αυτά που λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σε σχέση με την μορφή των ε, δαπανών. Το θέμα είναι μέχρι ποιο βαθμού ε, μπορεί κανείς να απλουστεύσει και παράλληλα να είναι σίγουρος ότι θα έχει πλήρη συμμόρφωση. Εγώ λοιπόν ε, πιστεύω ότι ως βουλευτές πρέπει να ακούμε και τις δύο πλευρές και εκείνους που αναζητούν τις ε, τις απαλλαγές. Από την άλλη όμως να ακούμε και τους πολίτες μας ε, που διαμαρτύρονται για τη γραφειοκρατία και για πολλά άλλα. Εμείς δηλαδή κάπως πρέπει να είμαστε στη μέση και να προσπαθούμε να ε, διαμεσολαβήσουμε. Όσον αφορά τους υπόλοιπους οργανισμούς υπάρχουν λίγα πράγματα που θέλω να πω. Έχω καταθέσει μία-δύο τροπολογίες αλλά σε γενικές γραμμές τα είπατε όλα. Είπατε όλα όσα έπρεπε να λεχθούν. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Η Κομισιόν δεν ξέρω αν επιθυμεί να παρέμβει. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να κάνω ε, κάποια σχόλια για το σχέδιο του ψηφίσματος. Πρώτα απ' όλα ε, θέλω να πω το εξής, ότι παρά τους ε, δημοσιονομικούς περιορισμούς, το επίπεδο των πληρωμών αυξήθηκε το 2012 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη έχει φτάσει ε, στα 11,6 νομίζω δισεκατομμύρια. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη και αυτό σημαίνει ότι έχουμε υπερεκτελέσει τον αρχικό προϋπολογισμό. Φτάσαμε στο 130% του προϋπολογισμού, κυρίως για τις ε, πληρωμές. Έχουμε την ε, μικροχρηματοδότηση. Αυτό είναι μια εξήγηση. Σε γενικές γραμμές η ε, εκτέλεση και όπως σας είπα το επίπεδο ε, χρηματοδότηση σε σχέση με προηγούμενα έτη είναι πολύ καλό. Σε σχέση με φέτος για τη Γενική Διεύθυνση της Απασχόλησης ε, έχουμε το 3,2% που είναι το λιγότερο από όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αύξηση σε σχέση με το 2011 που ήταν 2,2%. Δηλαδή ε, βρισκόμαστε κοντά σε αυτό το ποσοστό του 2011. Για να κατανοήσει κανείς την αύξηση είναι σημαντικό να επισημάνει ότι το 40% του συνόλου του ποσοστού σφάλματος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά ένα κράτος μέλος. Και για αυτό το κράτος μέλος η Κομισιόν στο ίδιο οικονομικό έτος ε, το 2011 εφάρμοσε ε, διορθώσεις 20%. Άρα το σφάλμα ήταν γνωστό και διορθώθηκε στο ίδιο οικονομικό έτος. Για καθαρά μεθοδολογικούς λόγους ε, αυτή η διόρθωση που είναι πολύ σημαντική δεν ελήφθη υπόψη στον υπολογισμό του σφάλματος και εάν αυτό είχε γίνει η κατάσταση θα ήταν σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τώρα τι μέτρα λάβαμε το 12 και το 2013. Πρώτα απ' όλα, συνεχίσαμε με την εφαρμογή της αυστηρής πολιτικής που είχαμε ακολουθήσει για πολλά χρόνια σχετικά με τη διακοπή ή αναστολή πληρωμών. Και ε, παρά αυτή την αυστηρή πολιτική κατορθώσαμε ε, να αυξηθεί λίγο όγκος των πληρωμών το 10 και το 11. Επίσης εφαρμόσαμε οικονομικές διορθώσεις το 2012 και επενδύσαμε σε αυτό που είπατε και είναι η απλούστευση. Πιστεύουμε ότι η απλούστευση είναι σημαντική ευκαιρία για να βελτιωθεί η λειτουργία του κοινωνικού ταμείου Γι' αυτό λοιπόν ε, την απλούστευση την εφαρμόσαμε σε όλα τα κρατημέλη, στα 24 από τα 28 προάγουμε την απλούστευση και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επόμενη περίοδο. Με βάση την αντίδραση που λάβαμε, θεωρούμε ότι οι προοπτικές προς την καλύτερη εφαρμογή της απλούστευσης ε, είναι υπαρκτές και θεωρούμε ότι θα υπάρξουν ε, θετικέ εξελίξεις όσον αφορά ε, τη λειτουργία και την εφαρμογή του Ταμείου. Αυτό που επίσης εφαρμόζουμε είναι οι καθαρές διορθώσεις ως μέσο. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στα κράτη-μέλη, τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με σημαντικές ελλείψεις στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με την Ευρώπη 2020, ε, οι ενέργειες αντικατοπτρίζουν στην πραγματικότητα πάνω από 50 εκατομμύρια άτομα συμμετείχαν από το 7 μέχρι το 11 και όσον αφορά ε, τα τελευταία στοιχεία πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν το 2011 συμπεριλαμβανομένων ε, περίπου 5 εκατομμυρίων νέων. Τώρα το 12 είχαμε 11 αιτήσει από τα κράτη-μέλη 259 εκατομμύρια και αυτό αφορούσε περίπου 10.000 εργαζόμενους και εκεί η ανεργία ήταν 42%. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι σε γενικές γραμμές παρότι υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτιώσεων τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Και το γεγονός ε, είναι ότι έχουμε ε, χαμηλό ποσοστό σφάλματος, αυτό μας καθησυχάζει. Όσον αφορά τους οργανισμούς, οι τέσσερις εκθέσεις είναι καλές, δεν τίθενται ε, πολλά θέματα. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό που παίζει ρόλο είναι ο χαρακτήρας των ε, προγραμμάτων. Τέλος, ε, πιστεύω ότι τα σχόλια που γίνονται από τους οργανισμούς, τις ετήσιες εκθέσεις τους, αφορούν ε, στην διαφάνεια και τις προσλήψεις. Merci beaucoup de, de ces précisions dont, dont nous tiendrons compte euh, dans... λάβουμε υπόψη της κυβερνήσεις και σας ευχαριστούμε. Κύριε Χαρκίν, σας ευχαριστούμε και εσάς. Ό,τι είπατε, ας γίνουν τροπολογία. Θα διευκρινιστούν όλα τα θέματα που είπατε. Μέχρι 7 Ιανουαρίου το μεσημέρι θα είναι η προθεσμία για την τροπολογια 22 22-23 Ιανουαρίου θα τη συζητήσουμε, 12 Φεβρουαρίου συμβαστικές και θα υποβληθούν μετά αυτά ή στην Ολομέλεια 17 Μαρτίου τελειώσει αυτό το σημείο της μεσής διατάξεως. Τώρα, φτάνουμε στο σημείο 26. Επ' αυτού θα δώσω το λόγο στην Edit Bauer αφορά τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο τη ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Voir euh, évoquer en négociation de manière relativement euh, sans trop de difficultés, en réalité se révèle être. Euh... Θεωρούσαμε ότι το ζήτημα θα είναι περίπλοκο και δύσκολο και, ε, και γι' αυτό και τελικά οι διαπραγματεύσει ήταν σκληρές. Thank you, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω καλά νέα. Ολοκληρώσαμε σήμερα το πρωί τις ε, διαπραγματεύσεις μετά από έξι ώρες διαπραγματεύσεων η ε, Κομισιόν και το Συμβούλιο ολοκλήρωσαν βέβαια κάτω από ορισμένε ε, προϋποθέσεις, κάποια προαπαιτούμενα, τα οποία που σε αυτή την περίπτωση μάλλον σημαίνει ότι ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις με την προϋπόθεση ότι το πακέτο επί του οποίου συμφωνήσαμε πρέπει να περιλαμβάνει το συντονισμό να υπάρχει δυνατότητα συλλογικών αποζημιώσεων, επίσης ε, να αντιμετωπίζεται η διακριτική μεταχείριση με βάση τον τόπο κατοικίας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι παρότι ο κανονισμός σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι σε μία συγκεκριμένη διάταξη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρει αυτό το πρόβλημα. Γνωρίζουμε όμως ότι ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν τη διακριτική μεταχείριση με βάση τον τόπο κατοικίας. Το Συμβούλιο αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτό το θέμα να ε, συμπεριληφθεί στο νομικό κείμενο. Έτσι λοιπόν Τελικά μπορέσαμε να καταλήξουμε ε, σε κάποια συμβαστική πρόταση, εφόσον πρόκειται για συμβασμό, δεν πρόκειται για τη βέλτιστη λύση, αλλά τέλος πάντων αποδεκτή είναι. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να περιμένουμε την ε, αντίδραση που θα υπάρξει μέχρι την Παρασκευή. Και εάν υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο, θα μπορούμε τότε να πούμε ότι πραγματικά Έχουμε μια εμπλουτισμένη πρόταση η οποία δεν προέκυψε με μεγάλη ευκολία, ήταν σκληρές οι διαπραγματεύσεις, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Ευχαριστούμε, συγκήτρια. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι. υπό την ηγεσία σας κινητοποιηθήκατε όλη η ομάδα των διαπραγματευτών για αυτό το κείμενο που αφορούσε την ελεύθερη ε, κυκλοφορία κατεξοχήν. Και επομένως στα πλαίσια αυτής θα έπρεπε να γίνουν σεβαστά τα κοινότητα των εργαζομένων. Έτσι με λίγα λόγια για να τα πούμε. Κλείσατε αυτό το συμβασμό και έτσι έχουμε αίσιο τέλος της διαπραγματεύσεις. Θα υπάρξει πάντως ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε τα αποτελέσματα όταν ξανεπιληφθεί η Κορεπέρ και εμείς ξανασυνεδριάσουμε. Τελειώσαμε το σημείο 26 και πάμε στο σημείο 27. 29-31 Οκτωβρίου 2013 είχαμε την προσωπία της Επιτροπής μας που μετέβη στην Αθήνα για να συναντήσει την ελληνική προεδρία. Θα πάει. Θα Πήγε 29-31 Οκτωβρίου. Και θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση γιατί θα σας υπενθυμίζω ότι σε αυτήν την προσωπία που πήγε στην Αθήνα 29-31 Οκτωβρίου είχαμε και τον Σέρκα, στην ε, Στάιμπρουκ, είναι Τσουμπέρ. Comme euh, euh, euh, locaux de l'État, si j'ose dire, Constantinos Poupakis et. Συνάντησε τον ε, κύριο Πουπάκη, ήταν η Σιλβάνα Ράπτη, την οποία συναντήσαμε και κατά την αποστολή, την αντιπροσωπεία εκεί επίση συναντήσαμε τους ε, ομολόγους μας, την Επιτροπή δηλαδή Επασχόλησης του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τους υπουργούς απασχόλησης οικονομικών, τον πληρωτή υπουργό για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ε, τον γενικό διευθυντή της διεθνής απασχόλησης, συζητήσαμε τα τις εγγύσεις για ε, τους νέους, τους κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους τους και πάρα πολύ σύντομα επισκεφθήκαμε ε, ένα πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους νέους να εργαστούν ε, πάνω στις νέες τεχνολογίες. Και αν θυμάμαι καλά, ε, πρόκειτο για εγκαταστάσεις, εργοστάσιο τέλο πάντων της Nokia. Nos activités, mais là en l'occurrence il s'agissait d'une activité euh, intéressante et qui permet... Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσπάθεια γιατί έτσι δίνει τη ευκαιρία στους νέους οι οποίοι παίρνουν δυσκολίε να βρουν με αυτή την προσφορά, της, ε, την προσπάθεια της εταιρείας να βρουν κάποια δουλειά. Θέλει κάποιος που έχει συμμετάσχει και κάποιος άλλος θέλει και να ρωτήσει κάτι βεβαίως και σας παραπέμπω στα Τώρα, έχουμε τώρα το θέμα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Το σημείο 27α αφορά τον κανονισμό για την έρευνα που θα αφορά την απασχόληση σε κοινότητες. Η Τατιάνα Ντανόκα έχει το λόγο γιατί είναι η δική μας συντάκτη. Η και να μας πει τι έγινε με τον τριμερή διάλογο που έγινε σήμερα το πρωί. Είναι ο δεύτερος ε, τριμερής διάλογος που έχει διεξαχθεί για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά υπό τη δική σας ε, καθοδήγηση και βέβαια και με την αρχική θέση της Επιτροπής. Είχαμε το δεύτερο τμήμα της έρευνας, το οποίο αφορά τα μοντέλα ad hoc και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα από ε, κατεξοδότηση πράξης. Βέβαια υπήρξαν κάποιες ε, συμβαστικές ε, προτάσεις από τον πρώτο τριμερή διάλογο και πολλοί πέμειναν ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή ε, πρέπει να έχουν περισσότερο λέγειν όσον αφορά το τον κατάλογο των ε, θεμάτων που είναι όμως πολιτικής σημασίας. Ε, πρέπει βέβαια να τα κοιτάξουμε όλα αυτά και πρέπει ε, να έχουμε κατά νου ότι οι ρυθμίσεις γίνονται τώρα με κατεξοδότηση πράξης. Δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε, όμως μετά από τον διάλογο το Συμβούλιο είπε ότι θα προτιμάσει τη συνάντηση της Κορεπέρ. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή. Και έχουμε το κείμενο το οποίο επαναλαμβάνεται βέβαια το κείμενο του ε, Κοινοβουλίου με κάποιες ε, αλλαγές. Ελπίζουμε ότι την ε, Παρασκευή όλα αυτά θα συμφωνηθούν ε, από το Συμβούλιο, αλλιώς δεν θα έχουμε ε, συμφωνία πρώτης ανάγνωσης. Και να αναφέρω και κάτι άλλο που αφορά στην συμφωνία μας. Υπάρχει η περίφημη δίτρα μη γνωμοδότησης. Αν δεν υπάρχει γνωμοδότηση, τότε η Επιτροπή δεν ε, θα εγκρίνει το σχέδιο εφαρμοστικών πράξεων. Τώρα η ε, πρόταση αυτή πρόκειται να αποσυρθεί. Ελπίζουμε λοιπόν ότι την Παρασκευή ε, το θέμα θα συμφωνηθεί στο Συμβούλιο και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Θα καταλάβατε όλοι πως πάλι και αυτό σχετίζεται με την επιτροπολογία. Και πάλι χρειάζεται το Κοινοβούλιο να επιμείνει για να δείξει πως δεν συντρέχει λόγος για να αλλάξουν οι λόγοι που χρησιμοποιήθηκαν ως νομική βάση για να εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις του συνθήκη και δεν υπάρχει λόγος τέλος πάντων να αναθεωρηθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου ως προς τις βασικές νομικές πράξεις. Μα τελικά επικράτησε η κοινή λογική μετά από μια αρκετά τεταμένη πρωινή συνεδρίαση. Ελπίζουμε ότι με τη γραπτή διαδικασία η Λιθωνική Προεδρία μέχρι την ε, Παρασκευή θα το έχει κλείσει το ζήτημα. Hm. Και εμεί ε, στην επόμενη συνεδρίασή μα σε αρχέ Ιανουαρίου θα επανέλθουμε για να το επιβεβαιώσουμε. Σα ευχαριστούμε ε, διότι δείξατε μεγάλη αποσίωση και φτάνουμε στο τελευταίο σημείο, δηλαδή απολογισμός ε, των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο ε, για την 96-71 οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και την παροχή υπηρεσιών. Η Δανούτα Νασνογεύσκα που είναι η συγγήτριά μας, ε, θα πάρει το λόγο για να κάνει απολογισμό των διαπραγματεύσεων. Δύο πρέσβεις ήταν παρόντες ε, ε, και για την Λιθουανική Προεδρία και για την επερχόμενη Ελληνική Προεδρία, αλλά και ο Επίτροπος ο αρμόδιος επίτροπος εκπροσώπησε την Επιτροπή. Παρακαλώ, jak państwo zapewne wiedzą dziewięć grudnia zostało przyjęte stanowisko przez radę do ε, ε, Πρόκειται για την ε, θέση του Συμβουλίου. Όπως είπατε λοιπόν κύριε Πρόεδρε, σήμερα είχαμε την πρώτη συνάντηση. Βέβαια ε, θα λέγαμε ότι πρόκειται περισσότερο για μια προκατακτική συνάντηση. Η πρόεδρος είπε ότι συμμετείχαν στη συνάντηση οι πρέσβεις της Λιθουανίας, άρα δηλαδή της απερχόμενης προεδρίας και ο πρέσβης της επερχόμενης προεδρίας, ο Έλληνας πρέσβης και συζήτησαν για τον τρόπο εργασίας. Επίσης ε, πήραμε και ένα ε, ημερολόγιο εργασιών. Εκεί προβλέπονται έξι συναντήσεις και προβλέπονται και για δύο περιττέρω συναντήσεις που ίσως κριθούν απαραίτητες. Έχουμε το άρθρο 9 και το 12, τα άρθρα 9 και 12 που είναι επίμαχα ε, άρθρα. Η θέση του Συμβουλίου εκεί είναι διαιρεμένη και επειδή οι εργασίες δεν είναι εύκολες, αποφασίσαμε οι εργασίες για τα άρθρα 1, 2, 4 και 5 το ένα είναι το subject matter, το δύο είναι οι ορισμοί, το τέσσερα είναι ο σύνδεσμος και το 5 αφορά την ενημέρωση. Στην ε, περίπτωση του άρθρου 5 ίσως ε, εκεί να συζητήσουμε κυρίως για την ε, πρόταση να διευρυνθούν περαιτέρω μεταφράσεις. Δηλαδή το Συμβούλιο δεν προβλέπει διευρυμένο σύστημα μεταφράσεων έτσι λοιπόν ε, προβλέπουμε να υπάρξει αργότερα και ε, να υπάρξουν εργασίε στο άρθρο 3 ε, που εκεί γίνεται λόγος για συγκεκριμένα στοιχεία πρόκειται για καταχρήσεις και αυταπάτες. Αυτά τα θέματα δεν ξέρω αν προκύπτουν αμέσως από τον τίτλο, την επικεφαλίδα του συγκεκριμένου σημείου. Γιατί ε, το Συμβούλιο έχει πρόβλημα με θέματα τα οποία δεν προβλέπονται στην αρχική του θέση. Έτσι λοιπόν η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρη. Σε αυτές τις ε, συναντήσεις ε, θα ασχοληθούμε και με το άρθρο 6, με το άρθρο 7 που είναι ο ρόλος των κρατών μελών. Θα θυμάστε ότι ε, έχουμε αλλάξει το άρθρο αυτό. Η πρόταση επιτροπής αφορούσε μόνο τις ε, υποχρεώσεις που έχουν σχέση με τη χώρα προέλευσης. και όσον αφορά τη συνεργασία και την απόσπαση των εργαζομένων θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι ε, στα κράτη υποδοχής. Αυτά όλα αφορούν το σύστημα ενημέρωσης για την εσωτερική αγορά στο άρθρο 3 οι διπραγματεύσει ε, θα είναι δύσκολες. Κατόπιν ε, θα είναι έντονες συζητήσει όσον αφορά το σύστημα ΙΜΗ. Το ε, Συμβούλιο προβλέπει ότι η συνεργασία πρέπει να είναι υποχρεωτική Ας δούμε λοιπόν και τις εργασίες για το τέταρτο κεφάλαιο. Πρόκειται για τον έλεγχο συμβατότητας με το άρθρο 9. Μετά άρθρο 10. Έλεγχη. Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά την εφαρμογή 11. Άρθρο 12. Αφορά τους δημόσιους διαγωνισμούς και αυτές οι συνεδριάσεις θα είναι πολύ πιο δύσκολες από ό,τι περιμέναμε. Γιατί το άρθρο 11 και το άρθρο 12 είναι ε, αντιφατικά <clears throat> άρθρα μεταξύ τους. Πάντως ε, θεωρούμε ότι στο Συμβούλιο τελικά ενδέχεται να επιτευχθεί η συμφωνία. και ελπίζουμε ότι θα ληφθεί μια απόφαση κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Κατά την έκτη τώρα συνεδρίαση θα γίνουν εργασίες για το έκτο κεφάλαιο, διασυνοριακή εφαρμογή και ούτω καθεξής, άρθρο 13 έως άρθρο 16. Και από το 17 μέχρι το 20 και το 23 και ίσως θα δούμε κατά πόσον θα υπάρξει κάτι για όλα αυτά τα άρθρα. Και στο, στην τελευταία συνεδρίαση ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες συζητήσεις για το άρθρο 13 όσον αφορά κυρίως τις κοινωνικές παροχές που είναι ένα θέμα ευαίσθητο για το Συμβούλιο. Άρθρο 14, τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εισάγει τη, τα θεμέλια για την απόρριψη ε, και εδώ ίσως ε, θα πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό λοιπόν το άρθρο, ε, αυτά είναι τα άρθρα που θα στηθούν. Ε, και ε, βεβαίως όλοι είναι ανοιχτοί για αλλαγές ή για συζητήσεις. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστούμε. Θα προσθέσω κι εγώ ένα σημείο. Για να είναι πληρέστερη η παρουσίασή σας, έχουμε γλωσσικό καθεστώς με τρεις γλώσσες, αγγλογαλλικά και πολωνικά προς το παρόν. Αλλά έχουν προβλεφθεί έξι τριμερείς εκ των οποίων κάποιοι ατελείωτοι, endless λέει αγγλιστή η Πρόεδρος, ε, όσο πάει. Το γλωσσικό καθεστώς, λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εξασφαλιστεί με το πέρας αυτής της ατελείωτης όσο πάει συνεδρίασης. Εξάλλου το Συμβούλιο τα, το βαρύ το πυροβολικό θα το ρίξει για, αυτά τα, για κάποια άρθρα. Στο πρώτο τριμερί που θα γίνει απουσία του πρέσβη, θα είναι αναπληρωτής, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση για τα 3, 9 και 12. Το Κοινοβούλιο προς το παρόν επιφυλάσσεται, δεν έχει τοποθετηθεί. Και ανάλογα με το πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις για το άρθρο 3, θα αποφασίσουμε ενδεχομένω να ε, αλλάξουμε τη σειρά διαπραγμάτευση των άρθρων, ούτως ώστε να ασχοληθούμε κατά προτεραιότητα με τα προβληματικά άρθρα. Αυτό θα είναι δυνατόν μόνο, μόνο εάν καταλήξουμε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα στη διαπραγμάτευση για το άρθρο 3. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο, θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια. Όχι, πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε και την μερίσια διάταξή μα. Ραντεβού στην επόμενη συνεδρίαση 9 Ιανουαρίου. Έκτακτη συνεδρίαση από τις 9 μέχρι τις 12.30. Αλλά μη φύγετε, μη φύγετε τελείως από, εδώ, από το κτίριο γιατί έξω είναι και ο Επίτροπος και θα πιούμε ένα ποτηράκι ε, για να γιορτάσουμε το τε, των εργασιών για το 2013 ήταν εξαιρετικά φορτωμένη χρονιά και το ξέρουμε, το νιώσαμε όλοι. Τα λέμε εδώ απ' έξω.